Buongiorno. Buongiorno. Così, in occasione della prima riunione. Eh... Λοιπόν, πρόκειται για την πρώτη πραγματική λειτουργική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ε, γι' αυτό και καθυστερήσαμε λίγο, αλλά έπρεπε να οργανωθούμε κάπως. Παίρνω αμέσως λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο σημείο είναι η αποδοχή των, της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, η πρόταση μπορεί να γίνει δεκτή. Έχω τώρα μία σειρά ανακοινώσεων εδώ. Η πρώτη αφορά τη διερμηνία. Έχουμε διερμηνία σήμερα σε 23 γλώσσες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σχετικά με την πολυγλωσία η οποία χαρακτηρίζει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσπαθήσουμε πάντα να έχουμε τις περισσότερες δυνατές γλώσσες στα, στα πλαίσια της, ε, των συνεδριασιών μας. Ανάλογα βέβαια και με την διαφυσιμότητα των διερμηνέων. Μερικές φορές θα πρέπει οι συνεδριάσεις μας να γίνονται σε αίθουσες τις οποίες δεν υπάρχουν ε, επαρκή δεν υπάρχει επαρκής αριθμός θαλαμίσκων και έτσι ε, θα υπάρχουν κάποιες γλώσσες λιγότερο. Ξέρετε επίσης ότι θα πρέπει να μειώσουμε το κόστος και γι' αυτό ζητώ από, όλους, ε, από όλα τα μέλη όταν δεν θα είναι παρόντες σε μια συνεδρίαση να ειδοποιούν την γραμματεία εγκαίρως έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε αν είναι δυνατόν τον αριθμό των γλωσσών στις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε. Οι e Γιατί στόχος όπως είπα είναι να μειώσουμε το κόστος της μετάφρασης και της διευμηνίας. Τώρα δεύτερον, η αναμετάδοση ε, η διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεών μας θα συνεχιστεί όπως εδώ και αρκετή, αρκετό καιρό. Να προσθέσω ότι όπως γνωρίζετε η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι η υπεύθυνη Επιτροπή για τη μείωση της χρήσης του χαρτιού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν ε, όσοι μετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και δεν θέλουν να παίρνουν χαρτιά με τα προγράμματα κτλ αλλά θέλουν να ενημερώνονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο που θα είναι έτσι κι αλλιώς διαθέσιμα όλα αυτά τα θέματα στην ιστοσελίδα μας. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να μην παίρνουν ε, σε χαρτί ε, τα τεκτενόμενα στην Επιτροπή μας να το δηλώσουν στη Γραμματεία. Τώρα, για αυτό το πακέτο καλωσορίσματος λοιπόν στην Επιτροπή μας θα το βρείτε μπροστά σας σε διάφορες γλώσσες και στη μητρική σας γλώσσα υποθέτω όλων ημών περιλαμβάνει μια εισαγωγή για τις εργασίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων με αρκετές πληροφορίες χρήσιμες για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με αρκετές άλλες δραστηριότητες για τις δραστηριότητες γενικότερα τις οποίες θα εμπλακούμε τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή αυτό το πακέτο στην σελίδα μας. Η επόμενη ανακοίνωση θα είναι ευχάριστη. Ως συνήθως, σήμερα το απόγευμα, 15 λεπτά πριν από την αρχή της απογευματινής συνεδριάσεώς μας, δηλαδή στις 14.45, θα κάνουμε την οικογενειακή μας φωτογραφία. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλα τα μέλη, παρακαλώ όλα τα μέλη να είναι παρόντες στις 3 παρατέταρτο εδώ, έτσι ώστε η φωτογραφία αυτή ε, να μπορέσει να ε, χρησιμοποιηθεί αργότερα. Εδώ θα γίνει η φωτογράφηση, στην αίθουσα στην οποία συνήθως θα συνεδριάζουμε. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα ε, γίνει την 3η Σεπτεμβρίου, το πρωί και το απόγευμα, στις 9 και στις 3. Η συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου ακυρώνεται. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα ε, στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Το επόμενο σημείο αφορά τις ε, ανακοινώσεις των συντονιστών. Στις 14 Ιουλίου στο Στρασβούργο συνεδρίασαν οι συντονιστές. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής έχουν αποσταλεί σε όλα τα μέλη και είναι πλέον διαθέσιμα ε, στους φακέλους σας. Δεν έχω λάβει παρατηρήσεις από πλευράς των συντονιστών και μπορεί να θεωρηθούν ε, δεκτά. Είναι στη διάθεσή σας πάντως, επαναλαμβάνω, και ε, με ηλεκτρονική μορφή. Νομίζω ότι τώρα περνάω στο τέταρτο σημείο της ημερησίας διάταξης στον προϋπολογισμό για το 2015. Ε, οι συντονιστές λόγω της εμπειρίας την οποία έχω σωρεύσει από το παρελθόν γιατί ήμουν γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου τα προηγούμενα χρόνια μου ζήτησαν να συντάξω εγώ τη γνωμοδότησή μας γιατί πρόκειται για γνωμοδότηση και την απέστειλα χθε ε, ηλεκτρονικά και μόνο στην αγγλική γλώσσα γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό θα ήθελα τώρα να αλλάξω το καπέλο μου και να μιλήσω σαν εισηγητής για τη γνωμοδότηση που συνέταξα ε, προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εγώ έχω στην ουσία υπογραμμίσει στην πρόταση που κάνω τις πιστώσεις ε, για τους τομείς που μας αφορούν στους επόμενους προϋπολογισμούς. Είναι υψηλότερες οι πιστώσεις υποχρεώσεων από τις πιστώσεις πληρωμών και αυτό ιστορικά θα έλεγα προκαλεί από χρόνο σε χρόνο την αύξηση των λεγόμενων ραλ αυτών των τμήματων δηλαδή των πιστώσεων που δεν ρευστοποιούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου που τρέχει ο προϋπολογισμός και που μένει να ρευστοποιηθούν τον επόμενο χρόνο. Εμείς έχουμε εντοπίσει τις θέσεις στον προϋπολογισμό, τις σχετικές ε, με τα θέματα που μας αφορούν είναι σαφές επίσης πως για ορισμένα προγράμματα υπάρχει κάποιος κίνδυνος λόγω της μείωσης των πιστώσεων πληρωμών σε ορισμένους τομείς. Στην γνωμοδότηση την οποία έχουμε συντάξει λέμε στο σημείο 7 ότι σχετικά με το πρόγραμμα LIFE σαν παράδειγμα και σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό έχουμε μεν μια αύξηση 23,3 εκατομμυρίων για το περιβάλλον και 7,2 εκατομμυρίων για τις κλιματικές αλλαγές. Ενώ όμως η αύξηση για το περιβάλλον θα έπρεπε να είναι επαρκής έτσι ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για το 2015. Το τμήμα το οποίο αφορά το περιβάλλον φαίνεται να αποδεικνύεται ανεπαρκές. Υπάρχουν ανεπαρκείς πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του 15. Αυτό σημαίνει ότι τον Οκτώβριο του 2015 θεωρητικά εξαντλούνται ε, οι διαθέσιμες πιστώσεις και αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή θα υπάρξει μια συγκεκριμένη έλλειψη πιστώσεων πληρωμών. Και γι' αυτό ζητάμε στη γνωμοδότησή μας από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν την επάρκεια των πόρων στην περίπτωση που χρειαστεί με διορθωτικούς προϋπολογισμούς, με συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτητα κρουαζιέρας θα έλεγα των εργασιών και των προγραμμάτων μας χωρίς να υπάρξουν στάσεις που συνδέονται και οφείλονται στις ελλείψεις πιστώσεων. Κάποια άλλα θέματα στα οποία έχουμε σταθεί και που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση αφορούν τις εξωτερικές υπηρεσίες. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ε, στον προϋπολογισμό των συνολικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έτσι ώστε να μειωθεί σε 5 χρόνια κατά 5% το προσωπικό των εξωτερικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μάλλον προβλήματα σε ορισμένες τέτοιες υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδιαίτερα σε αυτούς που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών προς τα έξω και που ε, χρηματοδοτούνται εν μέρη τουλάχιστον όχι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθείας αλλά ένα τμήμα των εσόδων τους προέρχονται από αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, επιχειρήσεις κτλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα θέσει μάλλον ένα κινδύνο τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών των οργανισμών καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν ε, σημειώσαμε ιδιαίτερα για δύο οργανισμούς το κρίσιμο της κατάστασης και ποια είναι τα προβλήματα τα οποία μπορεί να συνδεθούν με τη μείωση των πιστώσεων εις βάρος των ε, οργανισμών αυτών. Ταυτόχρονα έχουμε εμείς ε, επιμείνει στη σημασία που δίδουμε στις πιλωτικές και προπαρασκευαστικές δράσεις είναι προπαιδευτικές θα έλεγε κανείς ε, διαδικασίες ε, που προηγούνται των προγραμμάτων και υπάρχει ανάγκη τα πιλωτικά και τα προπαρασκευαστικά αυτά βήματα δράσης που συνδέονται με τη θεματολογία μας να χρηματοδοτηθούν πλήρως από τον προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν σε μια συνθετική γραμμή σας παρουσίασα ε, πάνω κάτω τη γνωμοδότηση θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αφρανσουά Καζανά και επίσης ε, τον Διευθυντή της ε, Διεύθυνσης για το Περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω μερικά λόγια για τον προϋπολογισμό για το περιβάλλον γενικότερα. Το ύψος των προβλέψεων είναι 480 εκατομμύρια για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015 και για τις πληρωμές λίγο λιγότερο από 400 εκατομμύρια, 380. Σε σύγκριση όλα αυτά με τον συνολικό προϋπολογισμό φαίνονται χαμηλά αυτά τα ποσά αλλά είναι μόνο το φανερό τμήμα του παγόβουνου. Πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι κλιματολογικές αλλαγές για να κινητοποιηθούν τα περιφερειακά ταμεία ή να χρηματοδοτηθεί η πολιτική εξωτερικών σχέσεων κλπ. Δεν έχουμε την ακριβή κατανομή των κοντιλίων αλλά περίπου 5% του κοινοτικού προϋπολογισμού αντιπροσωπεύουν όλα αυτά. Και εδώ και μερικά χρόνια αρχίσαμε να εφαρμόζουμε ένα σύστημα ίχνη λασιμότητας της χρήσης των κονδυλίων, ιδιαίτερα για την διατήρηση της βιοπικιλότητας. Ο προϋπολογισμός αυτός για το περιβάλλον κατά 80-85% είναι το πρόγραμμα LIFE και προγράμματα βοηθητικά άλλων οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είπε και ο πρόεδρός σας και τα πιλωτικά πειραματικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις. Για το 2015 οι προτάσεις μας ακολουθούν το, ΠολΔΙΠ, το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα και ό,τι προβλέπεται για τις δαπάνες των διαφόρων υπηρεσιών όπως του Ίδρυμα της Κοπενχάγης. Ακολουθούμε λοιπόν αυτά που επιβάλλει η δεοντολογία για, αυτές, για αυτού του είδους τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα. Για το 15 οργανισμούς. Για το 15 όπως είπε και ο πρόεδρος υπολογίζουμε ότι από τον Οκτώβριο αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις μας, μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στις πληρωμές και να χρειαστούν μεταφορές από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού. Δεύτερο θέμα για το 2015, η εισφορά μας στον οργανισμό για τα χημικά προϊόντα και ιδίως τα βιοκτώνα. ένα τμήμα των εισφορών αυτών προέρχεται από τα τέλη που επιβάλλουμε στις εταιρείε που εγγράφουν τα προϊόντα τους. Από το 11 έχει αρχίσει να γίνεται αυτή η εισφορά. Τώρα μειώθηκαν τα τέλη αυτά και το πρόβλημα θα γίνει πολύ σοβαρό το 2015 Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση πιο βιώσιμη για αυτό το πρόβλημα. Άλλο θέμα σημαντικό για το 2015 θα είναι η δεύτερη χρονιά εφαρμογής του πολιετούς δημοσιονομικού, αλλά στην ουσία για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί στην πράξη, θα στην πράξη οι συστάσεις του και το μεγαλύτερο τμήμα του προγράμματος LIFE και της διαχείρισής του έχει δοθεί σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό, ΕΑΣΜ λέγεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα χρησιμοποιηθούν και δημοσιονομικά εργαλεία νέου τύπου για πρώτη φορά διαχειριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών ή για την βιοπικιλότητα. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που ήθελα να σας πω. Ίσως τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου εδώ, κλερκ, για να προσθέσει μερικά. Ευχαριστώ. Για τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και την ευημερία των ζώων και των φυτών, τα συνολικά ποσά είναι περίπου 475 εκατομμύρια σε προβλέψεις και κατανέμονται ανάμεσα στη δημόσια υγεία και την ευημερία φυτών και ζώων και υπάρχουν τρεις οργανισμοί, η ΕΦΣΑ, η μάρκεο ΕΦΣΕ, που τα διαχειρίζονται. Τα ποσά αυτά ανταποκρίνονται στο δεύτερο έτος του πολιετούς προγράμματος που είχε εγκριθεί και για τους τρεις αυτούς οργανισμούς που ανέφερα οι πληρωμές τους ανταποκρίνονται στα ποσά που προβλέφθηκαν από τον Ιούλιο 13. Για τις δε πληρωμές περίπου τα ίδια ισχύουν με αυτά που είπε ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών. Υπάρχει δηλαδή μια μείωση λόγω του των δημοσιονομικών προοπτικών και στο τέλος του έτους θα υπάρξουν ορισμένα προβλήματα πληρωμών, αλλά αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από, το ακριβές, από την ακριβή χρονική στιγμή που θα αρχίσει να εφαρμόζεται και να εκτελείται ο προϋπολογισμός. Πρέπει να δούμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή κατά τη χρήση του προϋπολογισμού πώς θα είναι τα πράγματα. Οι διακανονιστικοί οργανισμοί που σας ανέφερα για το προσωπικό τους τουλάχιστον ε, και τι έχουν πληγεί από αλλά μπορούμε να κάνουμε μια ανακατανομή μεταξύ τους του 1% του προσωπικού και αυτό θα ισχύσει και για τους τρεις αυτούς οργανισμούς, ΕΝΤΕΣΕ, και ΕΜΑ. Αυτά. Ευχαριστώ. Yes, thank you, Chair. Ο κύριος Βουίτεμα, ευχαριστώ και Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση που έχετε συντάξει και σας συγχαίρω. Δύο λόγια τώρα και για τα όσα είπατε εσείς και για τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κενό αυτό μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Είναι σημαντικό να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει το χάσμα αυτό για τους οργανισμούς Χαίρομαι που ενισχύεται ο ρόλος του εκτελεστικού οργανισμού για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις που θα βοηθήσει να ενισχυθεί το επιχειρήν και να ληφθούν υπόψη και προβλήματα του περιβάλλοντος, αλλά και να διατηρηθεί ο πρωτοπόρος ρόλος των βιομηχανιών μας στην πράσινη οικονομία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα βοηθήσει στην παραγωγή νέων προϊόντων. Τώρα για την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, της ε, προστασίας των καταναλωτών, ε, της υγείας μάλλον, εδώ με ανησυχεί η έλλειψη χρηματοδότησης για κολλητικές ζωονόσους, για τον αυτόν πυρετό των χείρων, που το κόστος του και μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και εμείς στο αποθεματικό έχουμε μόνο 400 εκατομμύρια. Αυτά ήταν με λίγα λόγια τα όσα ήθελα να σημειώσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς κύριε Γκρότε. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια που σε λιγότερο από μια εβδομάδα προλάβατε και συντάξατε την γνωμοδότηση. Ακούσαμε πάλι για τους οργανισμούς, ότι δηλαδή για τους οργανισμούς πάλι κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή τους φορτώνουμε όλο και περισσότερα καθήκοντα χωρίς να εξασφαλίζουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και περικόπτουμε και το προσωπικό τους. Αυτό το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη παλαιότερα εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και με τη βοήθεια της Γιούτα Χάουκ που ήταν τότε η διαρκή συζήτρια. Στο μέλλον πρέπει να πάρουμε τα πράγματα αυτά σοβαρότερα υπόψη γιατί έχουμε πολύ καλή επαφή με τους οργανισμούς και μας θέτουν διαρκώς υπόψη το ίδιο θέμα, ότι οι απαιτήσει μας απέχουν πολύ από την χρηματοδότηση που τους εξασφαλίζουμε. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί με πιο εύκαμπτο τρόπο και κυρίως να χαρίσουμε προσοχή στα όσα λένε και για τους διάφορους οργανισμούς όπου εισπράττουν και τέλη για την καταχώρηση προϊόντων. Βέβαια για το ύψος των τελών μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά έχει σημασία ο προϋπολογισμός τους να είναι εξασφαλισμένος. Σας ευχαριστώ, Γκεμπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου σας συγχαίρω για την πρώτη σας αυτή εισήγηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δύο ερωτήσεις τώρα που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό και θα ήθελα να έχω κάποια απάντηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, για την βιοπικιλότητα. Στη βάση της ίδιας της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είδα ότι η Επιτροπή υπολογίζει ότι χρειαζόμαστε περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για να καλύψουμε τους στόχους μας. Εγώ έχω καταθέσει ορισμένες γραπτές ερωτήσεις, το έκανα αυτό λίγο πριν από την πάυση για τις εκλογές, και οι απαντήσεις που έλαβα με εξέπληξαν. Εγώ δεν αναφερόμουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που είναι διαφανής και ξεκάθαρος, αλλά για τους προϋπολογισμούς των χωρών μελών που χορηγούνται για τη βιοπικιλότητα. Και η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Δεν έχει ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι διαθέτουν στου εθνικού του προπολογισμού οι χώρε μέλη για τη βιοπικιλότητα. Η ερώτησή μου λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ποιο είναι το επόμενο τη βήμα. Πώ θα επιτύχουμε το, του στόχου τη στρατηγική μα για τη βιοπικιλότητα, γιατί με 3,46 δισεκατομμύρια στο πρόγραμμα LIFE κατεσπαρμένα σε 7 χρόνια, δεν φτάνουν για τίποτα. Δεν φτάνουν ασφαλώς ούτε για ένα χρόνο. Θα αναλάβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλη την ευθύνη για τη βιοπικιλότητα αφαιρώντας την από τις χώρες μέλη. Τι πρόκειται να κάνει για να ασκήσει περισσότερη πίεση στις χώρες μέλη έτσι ώστε να κάνουν πιο διαφανείς τους προϋπολογισμούς τους για τη βιοπικιλότητα. Και η δεύτερη ερώτησή μου αναφέρεται στη βιοπικιλότητα και πρόκειται για το αγροτικό περιβάλλον. Πέρσι μαζί με την ομάδα των φιλελευθέρων κατέθεσα προϋπολογισμούς, στο, ε, ε, κατέθεσα τροποποίηση συγγνώμη, στον προϋπολογισμό για να μπει ένα μέρος του σχετικού προϋπολογισμού στο αποθεματικό. Διότι έχουμε για τα προγράμματα Agri Environment, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο είναι το ποσόν, νομίζω ότι είναι και αυτό πάλι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια και εάν το συγκρίνετε με τον επταετή προϋπολογισμό του προγράμματος Life θα δείτε τι μεγάλη διαφορά έχει. Σύμφωνα όμως με το ελεγκτικό συνέδριο οι ευεργετικές επιπτώσεις των περιβάλλων αυτών των 2,5 δισεκατομμυρίων είναι απολύτως άγνωστες. Ίσως είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αυτό που ήθελα πέρσι με τις τροπολογίες αυτές στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι να βάλω 10% του προϋπολογισμού Agri Environment στο αποθεματικό και να διατεθούν τα χρήματα αυτά μόνον όταν θα έχουν αποδειχτεί οι ευεργετικέ επιπτώσει στο περιβάλλον του προπολογισμού αυτού, είτε από τι χώρε μέλη είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιε εξελίξει υπήρξαν από πέρσι, διότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να ξοδέψουμε τόσα πολλά χρήματα σε κάτι που έχει τόσο λίγε επιπτώσει για του στόχου του προπολογισμού, όπω αυτό το πρόγραμμα Agri Environment. Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ για τη διοργάνωση τόσο σύντομα αυτής της συνάντησης. Βέβαια δεν μπορώ να τα δω όλα λεπτομερώς, αλλά θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Πρώτον, νομίζω ότι κάπου πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι κυβερνήσεις των χωρών μελών είναι υποπίεση να μειώσουν τους προϋπολογισμούς τους και τις δαπάνες τους. Πολλές φορές τη αιτήσει και με αποπίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Δεν μπορούμε νομίζω να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του περιβάλλοντος πρέπει να στηρίζεται σε τέτοιες αρχές συστηματικών περικοπών, αλλά αυτό ισχύει για όλα τα τμήματα βέβαια του προπολογισμού. Πάντως νομίζω ότι θα ήθελα να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πειθαρχία και αυστηρότητα αντί από απλή συστηματική περικοπή. Οι μορισμένα παράγοντες που πρέπει να προστατευτούν να προστατεύονται και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν θέματα που είναι χαμηλότερης προτεραιότητας γιατί το θέμα δεν είναι απλώς ότι στιβάζουμε συνεχώς δαπάνες, είναι ότι έχουμε προτεραιότητες που πρέπει να τις εφαρμόσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε. Λένε ότι τα καλύτερα μέτρα είναι αυτά που είναι δημοσιονομικό ουδέτερα, δηλαδή δεν ε, αυξάνουν τις δαπάνες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο πειθαρχημένοι, να ξέρουμε δηλαδή γιατί αυτός ο κανόνας του δημοσιονομικού σου δετέρου δεν μπορεί πια να εφαρμοστεί και χρειάζονται περισσότερα χρήματα για ορισμένα θέματα. Αν συνεχίσουμε απλώς να στηβάζουμε όλο και περισσότερα καθήκοντα στους οργανισμούς δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα καθήκοντά τους. Ίσως να μπορούν οι οργανισμοί αυτοί να πραγματοποιήσουν και περισσότερες εξοικονομήσεις, αλλά πρέπει αυτό να το εξετάσουμε με τις περικοπές που προτείνονται του προσωπικού ή της ανακατατάξης. Θα κατοθέσουμε λοιπόν ορισμένες τροπολογίες, αλλά σας ευχαριστώ γενικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ούτως ή άλλως αναλάβει διεθνώς πολλές υποχρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Και τώρα άκουσα πριν από ένα μήνα ότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες χρηματοδοτικά να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει διεθνώς. Μήπως μπορεί να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πρόεδρε να επανέλθω στο θέμα των οργανισμών που γνωρίζω πρόκειται για την υπηρεσία φαρμάκων του Λονδίνου. Εδώ και χρόνια του δίδουμε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, ευθύνες, βαρύτατες. Είναι πολύ σημαντική η λειτουργία του οργανισμού αυτού. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να του τις αφαιρέσουμε. Πρόκειται για την πρόληψη στον τομέα της φαρμακολογίας για τις αδειοδοτήσεις ε, νέων φαρμάκων και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ορισμένα φάρμακα, σκευάσματα καινοτόμα, τα οποία θα πρέπει να περάσουν από μια αδειοδότηση κυκλοφορίας ε, της ευρωπαϊκής αυτής υπηρεσίας. Συνεπώς λοιπόν ε, κάθε χρόνο πρέπει να δίνουμε μάχη στον προϋπολογισμό έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ο οργανισμός αυτός θα έχει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε επίσης ότι επιβαρύνουμε τις εργασίες της υπηρεσίας, του ζητάμε επίσης να λειτουργεί και πιο γρήγορα και μειώνουμε τις πιστώσεις. Δεν ξέρω, ίσως κάποιους οργανισμούς κάτι να μπορούμε να κάνουμε με μείωση, αλλά όχι στον οργανισμό για τα φάρμακα. Πρέπει λοιπόν ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένου οργανισμού να επιτρέψει να διασφαλίσουμε για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη βέλτιστη δημόσια υγεία και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των σκευασμάτων. Ευχαριστώ. Εκχάουτ, κύριος Εκχάουτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ για τη γνωμοδότηση σας. Παρόμοια ερώτηση παλαιότερα όταν η Γιούτα Χάουκαν ελάμβανε όλα αυτά, ένα από τα πράγματα που έκανε ήταν να αποκαταστήσει τα, τους αριθμούς, τα ποσά δηλαδή, του σχεδίου του προϋπολογισμού. Η ερώτησή μου προς εσάς κύριε Σιγητά, προτίθεστε να το πράξετε αυτό ή αναμένετε να το κάνουν τα μέλη μέσω τροπολογιών. Λοιπόν δεν υπάρχουν άλλοι. Θα δώσω κάποιες απαντήσεις και μετά θα ζητήσω επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει. Είναι σαφές ότι όπως πάντα έχουμε κάνει η πρόταση ε, προϋπολογισμού την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πιστώσεις και πληρωμές, πιστώσεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. Ε, πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι πιστώσεις πληρωμών από πλευρά του Συμβουλίου ε, κουρεύονται για να μείνουμε μέσα σε μια συνολικότερη δαπάνη. Μια γενική γραμμική θα έλεγα διαδικασία που δεν λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους ανάγκες, απλά θέλει να μειώσει το συνολικό ποσό. Η πρόβλεψη την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σωστά σταθμισμένη και λαμβάνει υπόψη τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται και στους οργανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα προγράμματά του. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα παρουσιάσω και θα καταθέσω όλες τις τροπολογίες έτσι ώστε να προσπαθήσω να αποκαταστήσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Προϋπολογισμού με τη σειρά της θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε στα πλαίσια της ε, διαβούλευσης κάπου. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει κάποιες απαντήσεις στους τομείς αρμοδιότητάς της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα δύο ερωτήματα που τέθηκαν προς την Επιτροπή για τη Βιοπικιλότητα και τα περιβαλλοντικά. Για τη βιοπικιλότητα και το κρυμμένο μέρος του παγόβουνου που έλεγα πριν, η Κομισιόν θα αποτελέσει υπόδειγμα, θα δώσει το καλό παράδειγμα μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος ανείχνευσης ή χνηλασιμότητας των δαπανών και της χρήσης τους. Για τον προπολογισμό των χωρών μελών, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν με βάση αυτά που πρότεινε το Ελεκτικό συνέδριο για τη Βιοποικιλότητα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας αναφέρουν τι δαπάνες εφαρμόζουν για αυτόν τον σκοπό και έτσι να καταλήξουμε σε κάποια, κάποιο συντονισμό ή συνέπεια αυτών των ε, εκθέσεων. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ως προς τα μέτρα για το περιβάλλον θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι καλό ότι προς την πρόσφατη αξιολόγηση αποτίμηση των δαπανών του προϋπολογισμού με κριτήριο την νομιμότητά τους καθώς και την αποτελεσματικότητά τους το ελεγκτικό συνέδριο γράφει συνεχώς όλο και περισσότερες ειδικευμένε εκθέσεις για τύπους μέτρων. Το έχει κάνει για τη βιοπικιλότητα και για τη χρήση του νερού στην κοινή αγροτική πολιτική ή για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Αν και λοιπόν δεν συμφωνούμε πάντοτε με το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει, προβλέπεται ένας μηχανισμός, μια διαδικασία επίλυσης διαφορών οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα εξεταστούν δεόντως και θα δούμε κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικές. Θα υποβάλουμε τα συμπαράσματα αυτά και στο Κοινοβούλιο. Για τις κλιματολογικές αλλαγές θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο μου Βανόριμπεκ. Σας ευχαριστώ και εσάς και τον Πρόεδρο. Υπάρχουν πέντε διεθνείς συμβάσεις στις οποίες συμμετέχουμε για την αντιμετώπιση των κλιματολικών αλλαγών. Η μία είναι του ΟΗΕ, υπάρχει το πρωτόκολλο του Κιώτο, υπάρχει το θέμα των πληρωμών για τις εκπομπές διοξιδίου, υπάρχει το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ που προστατεύει τη ζώνη του όζοντος Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου 850.000 όσοι, να το πω έτσι, τέλη που πληρώνουμε το χρόνο. Και είναι βέβαιο, έχει επιτευχθεί ότι θα μπορέσουμε να τα πληρώσουμε αυτά και φέτος και του χρόνου. για να απαντήσω για τον αυθόδη, για τον πυρετό των χείρων. Το δημοσιονομικό πλαίσιο που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουνίου και άρχισε να εφαρμόζεται από τις 30, καθορίζει τους κανόνες και το κόστος για την εξάλληψη των επιζωτιών τέτοιου είδους. Είναι ένα, υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησής τους και υπάρχει κατάλογος των αναγνωρισμένων επιζωοτιών. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Θα πρέπει να σας θυμίσω τώρα τις προθεσμίες. Όπως γνωρίζετε φέτος η διαδικασία του προϋπολογισμού είναι πολύ πιο σύντομη, μιας και ήταν μια εκλογική χρονιά και οι χρόνοι που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένη προθεσμία για την κατεύθυνση προϋπολογισμών, ε, τροπολογιών στον προϋπολογισμό είναι 24 Ιουλίου, αύριο 16 απογευματινή. Όπως και η προθεσμία επίσης για τις ε, τροπολογίες στην γνωμοδότηση, τροπολογίες που θα πρέπει να είναι ε, διατυπωμένες μόνο στην αγγλική γλώσσα. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τη συνεδρίασή μας την 3η Σεπτεμβρίου. Το μοναδικό που θα ήθελα εδώ να προσθέσω είναι πως όλες οι προτάσεις για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικέ δράσεις θα πρέπει να παρουσιαστούν υπό τη μορφή τροπολογιών μέχρι αύριο το απόγευμα πάλι ε, στις 4. Λοιπόν δεν έχω κάτι άλλο εδώ, περνώ στο επόμενο θέμα της μέρης διάταξης. Παρασκευαστικές εργασίες για τη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα το Σεπτέμβριο του 2014. Όπως γνωρίζετε, στις 23 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Μπαν Κιμούν, θα οργανώσει μια διάσκεψη κορυφής παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση κορυφής αυτής έχει σαν στόχο να κινητοποιήσει τις πολιτικές δυνάμεις στα πλαίσια της διάσκεψης για το κλίμα που θα γίνει στη Λίμα και στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2014 ε, και του 2015. Ο Γενικός Γραμματέας Μπαν Κιμούν λοιπόν έχει προσκαλέσει κυβερνήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να κάνουν προτάσεις στη συνάντηση κορυφής έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιδιώξουμε και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών. Έχουμε εδώ τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης ε, Κλιματολογικών Αλλαγών, Τζόστε Μπέικερ, που θα μας παρουσιάσει το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι εργασίες προετοιμάζοντας τη συνάντηση κορυφής, τη διάσκεψη κορυφής. Και θα είναι στη διάθεσή σας αν θέλετε να θέσετε και κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, 10 με 15 λεπτά παρακαλώ. Έχει το λόγο ο Τζος Τελμπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για μένα είναι μεγάλη χαρά η παρουσία μου εδώ στην Επιτροπή σας, υπό την Προεδρία σας. Είναι πολύ σημαντική η Επιτροπή και η δράση της στο παρελθόν είναι εντυπωσιακή. Ήταν εντυπωσιακή. Το ίδιο αναμένουμε λοιπόν και για το μέλλον. Να περιοριστώ σε δύο-τρία θέματα για τη διάσκεψη Ban Το σημαντικότερο είναι ποια είναι η σημασία της στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Θα είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών εδώ και πολλά χρόνια για να προετοιμαστεί η συμφωνία των Παρισίων για τις κλιματολογικές αλλαγές το 2015. Τι θα συζητηθεί λοιπόν στη διάσκεψη Ban Θα είναι πολύ σημαντικό για την προετοιμασία αυτή. Θα σας πω μερικά λόγια ως προς το που βρισκόμαστε για με αυτή τη Διεθνή Κλιματολογική Συμφωνία. Οι επιστήμονες συλλογικά εκφραζόμενοι στην έκθεση IPCC είπαν ότι αν δεν ελεγχθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου στο τέλος του αιώνα θα αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 2,6 με 4,8 βαθμούς. Πρέπει λοιπόν να αποφευχθεί αυτό πάση θυσία και χρειάζεται μια σφαιρική κλιματολογική συμφωνία για να μειωθεί η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας σε κάτω από δύο βαθμούς. Όπως είχε ήδη συμφωνηθεί εξάλλου και στα πλαίσια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τις κλιματολογικές αλλαγές. Το 11 λοιπόν συμφωνήθηκε να προετοιμαστεί μια νέα σφαιρική συμφωνία μέχρι το 2015 για να περιοριστεί ακριβώς αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας σε δύο βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ σημαντικό για μας αλλά και για πολλά άλλα κράτη εκτός Ένωσης ότι για πρώτη φορά η συμφωνία αυτή θα εφαρμόζεται σε όλους τους συμβαλωμένους και όχι μόνο στους λεγόμενους της προσθήκης 1 του παραρτήματος 1 γιατί ο κατάλογος εκείνος είναι από το 92. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο στόχος πρέπει η Ένωση να συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο πιέζοντας για αυστηρά μέτρα για όλες για τις περισσότερο σημαντικές οικονομίες του κόσμου. Πέρυσι στη Βαρσοβία συμφωνήθηκε οι κύριες οικονομίες να υποβάλουν τις συνεισφορές τους, τα προτάσεις τους σε 8 μήνες από τότε για να γίνει μια αξιολόγηση του στόχου αυτού κάτω των 2 βαθμών Κελσίου πριν από την τελική συμφωνία το Δεκέμβριο του 2015 στο Παρίσι. Η Ένωση θα εφαρμόσει το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ήδη συζητιούνται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης οι προτάσεις μέχρι τον Οκτώβριο φέτος. Επίσης ενθαρρυντικά νέα έρχονται και από τη ΣΥΠΑ και επίσης ενθαρρυντικά από την Κίνα που συζητάει μια πιθανή, ένα πιθανό καθορισμό ημερομηνία για τον περιορισμό των εκπομπών. Άλλε χώρε όπω η Ιαπωνία, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, ο Καναδά, η Αυστραλία και άλλε δεν έχουν ακόμη επικυρώσει ότι θα υποβάλουν προτάσει μέχρι το τέλο του 2015 εγκαίρω. Αυτή είναι η σημασία που έχει η διάσκεψη του, γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους αρχηγούς κρατών με θέμα τις κλιματολογικές αλλαγές. Στην Λίμα 12 μήνες πριν, το Δεκέμβριο φέτος δηλαδή, 12 μήνες πριν τη διάσκεψη των Παρισίων θα γίνει μια τελευταία αξιολόγηση δεν είναι η ίδια διάσκεψη με τη διάσκεψη που λέγεται Ban Ki-moon, αλλά θα έχει και αυτή μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό ρόλο και ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τους αρχηγούς των κρατών να πάνε στη Λίμα και να τολμήσουν να κάνουν θαραλέες προτάσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλοι οι κύριες οικονομίες του κόσμου πρέπει να αποδείξουν ότι δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2015 και οι πτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες να τύχουν κάποια διασφάλισης ότι θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν ανάλογα μέτρα. Ο Βέβαιος Μπαρόσο θα εκπροσωπήσει την Ένωση και πολλοί αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, ο Επίτροπος Χέντεγκαρτ και πολλοί υπουργοί περιβάλλοντος επίσης θα πάνε στη Νέα Υόρκη για να συνεννοηθούν. Πάνω από 100 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων θα παραστούν και της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας, του Μεξικού που έχουν ήδη επικυρώσει ότι θα πάνε και φαίνεται ότι και ο πρόεδρος Ομπάμα θα συμμετάσχει. Η Ένωση λοιπόν πρέπει και αυτή να εκπροσωπηθεί δεόντως από τους αρχηγούς κρατών για να δείξουν ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν κάτι για τις κλιματολογικές αλλαγές. Τι θέλει λοιπόν να πετύχει η Ένωση στην διάσκεψη αυτή. Το σημαντικότερο θέμα θα ήταν οι ηγέτες του κόσμου να επαναλάβουν τη δέσμευσή τους να υπάρξει συμφωνία στο Παρίσι. Τέτοια που να οδηγεί σε μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου. Ο στόχος του 2030 θα καθοριστεί, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές ήδη του 2015, όπως είχαμε πει και στη Βαρσοβία. Πρέπει λοιπόν η Ένωση επίσης να αποδείξει, να δείξει ότι η δεσμεύση μας για το 2020 δεν αφορούν μόνο την Ένωση αλλά είναι διεθνείς στόχοι και ότι μάλλον θα ξεπεράσουμε και τους στόχους του 2020. Σήμερα σχεδόν τους έχουμε πετύχει αυτούς τους στόχους του 20, γιατί μειώσαμε τις εκπομπές μας κατά 18% ενώ ο στόχος ήταν 20%. Επίσης ελπίζουμε να δημιουργήσουμε εταιρικές σχέσεις και συμμαχίες και με άλλες χώρες γιατί πολλά από τα χρήματα που δαπανούμε για προγράμματα συνεργασίας αφορούν και την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Η διάσκεψη πρέπει να δείξει ότι υπάρχει πολιτική συνένεση και θέληση προσαρμογής ιδιαίτερα για τις πτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες. Εξάλλου η Ένωση σκοπεύει επίσης να επαναλάβει τη δέσμευσή της ότι θα διασφαλίσει την πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια για όλους μέχρι το 2030 δεσμευόμενη για σφαιρική προοδευτική μείωση των αερίων θερμοκηπίου σε και την υποκατάσταση ορυκτών πηγών ενεργείας από ανανεώσιμες. Μετά τη διάσκεψη Μπανκιμούν θα προετοιμαστούν οι διαπραγματεύσεις στη Λίμα το Δεκέμβριο φέτος και γι' αυτό φαντάζομαι ότι πολλοί ηγέτες θα αναφέρουν τι πρέπει να γίνει όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και τι πρέπει να κάνουν οι διαπραγματευτές μας στη Λίμα. Από όσο ξέρουμε θεωρούμε ότι καιρός είναι στη Λίμα να ακουστούν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια πρόταση για την μείωση, διαφάνεια, χρηματοδότηση, αξιολόγηση και άλλα σημαντικά στοιχεία αντιμετώπιση των κλιματολογικών λόγων. Επίσης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια απόφαση για το εύρος των ε, χρηματοδοτήσεων που σκοπεύουν να χορηγήσουν διάφορες χώρες Στη Λίμα πρέπει επίσης να ακουστούν διακανονισμοί για τη διεθνή διαδικασία που θα αναλύσει τις προτινόμενες συμβολές και ποσά πριν από το Παρίσι. Αυτές οι προτινόμενες εισφορές Συγχωρείτε γιατί εδώ έχει όλο αρχικά και δεν τα ξέρω. INDC το λέει αυτό, τις προτινόμενες συμβολές. Για να μειωθούν οι εκπομπές και αυτό θα ήταν το σημαντικότερο στοιχείο των διαπραγματεύσεων. Τι θα γίνει για να μειωθούν οι εκπομπές, περιορισμός τους. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με την προσαρμογή και τη χρηματοδότηση όλων αυτών. Τέλος για τη χρηματοδότηση αυτή στη Λίμα πρέπει να γίνει μια απτή πρόοδος για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών, ιδιαίτερα για το θέμα της εκμετάλλευσης του λεγόμενου πράσινου ταμείου. Στη διάσκεψη Ban Ki-moon λοιπόν πρέπει να δοθεί μια νέα ορμή για τις διαπραγματεύσεις αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών, ιδιαίτερα εν ώψη του των Παρισίων 2015. Και το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο βήμα προς τη διάσκεψη αυτή θα είναι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων στη Λίμα φέτος. Και με αυτή τη βάση νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος, προς την κατεύθυνση αυτής της σφαιρικής συμφωνίας στην οποία σκοπεύουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει αρκετοί συνάδελφοι το λόγο. Ο κύριος Λίζε θα είναι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Γενική Διευθυντά. Θα ήθελα πρώτα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να τονίσω ότι βρίσκω σημαντικό αυτό που είπατε ότι όλες οι χώρες που παράγουν σημαντικά, σημαντικά ποσά εκπομπών θα πρέπει να κάνουν την ίδια προσπάθεια. Είναι σημαντική αυτή η αρχή που επιτεύχθηκε τώρα και που πρόκειται ή μάλλον πρέπει να επικυρωθεί στο Παρίσι. Πρέπει τώρα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο για τη σχέση Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται ότι στην Κίνα η τιμή του τόνου διοξιδίου του άνθρακος είναι διπλάσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να με εξηγήσετε και τα σχέδια των ΗΠΑ τώρα για τον περιορισμό των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Σε όλα αυτά τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν ως στόχο ιδίω την βιομηχανία η οποία παράγει αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να εξετάσουμε και το λεγόμενο carbon leakage, τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών δηλαδή σε περιοχές όπου είναι οι όροι ευνοϊκότεροι για αυτές από άποψη εκπομπών. Πρέπει να δώσουμε όθηση σε καινοτομίες. Επίσης θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε με την κύρωση της δεύτερης φάσης υποχρεώσεων του Κιώτο. Δεν είναι ικανοποιητικά τα όσα γνωρίζουμε από εκεί, διότι στην ουσία συμμετέχει μοναχά η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει εμείς οι ίδιοι, αυτοβούλος, το 20% μείωση δηλαδή μέχρι το 2020. Και είναι σημαντικό για τη διεθνή αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να έχει ολοκληρωθεί και επικυρωθεί η προσπάθεια αυτή μέχρι το Παρίσι. Επίσης ένα επίκαιρο θέμα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τη στρατηγική της για το 2030 διότι μέχρι τώρα έλειπε κάτι από τη στρατηγική αυτή σχετικά με την αποδοτικότητα της χρήσης της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι μάθαμε και μας ανησύχησε αυτό, θα ζητήσει μόνο 25% αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας μέχρι το 2030. Το κοινοβούλιο έχει ζητήσει 40%. Εγώ είμαι ρεαλιστής και είμαι βέβαιος σχεδόν ότι τα 40% δεν θα επιτευχθούν. Αλλά θα ήθελα τουλάχιστον η Επιτροπή σήμερα να εγκρίνει μια τιμή, ένα όριο δηλαδή, που να είναι σαφώς άνω του 25%. Διότι η αύξηση αποδοτικότητας της χρήση της ενέργειας είναι από τους πιο οικονομικούς τρόπους για την επίτευξη των στόχων που έχουμε βάλει για τη μείωση των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Και στο κάτω της γραφής το ηλεκτρικό ρεύμα που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε, τόσο το καλύτερο. Δεν έχει καμιά ανάγκη ούτε από αυξημένες επενδύσεις, ούτε τίποτε άλλο σχετικό. Καλύτερα λοιπόν να διαθέσουμε τους πόρους σε αυτά, στην βελτίωση της χρήσης της ενέργειας, στην καλύτερη μόνωση των κτηριών μας και ούτω καθεξής. Αυτά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 was wir ja jetzt schon fast erreicht haben. Wir sind bei 19 äh, Έχουμε σχεδόν επιτύχει μέχρι τώρα, ήδη από το 2014, στο δρόμο προς το Παρίσι πρέπει ακόμα να κάνουμε μια προσπάθεια. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και θα κάνουμε περισσότερα. Να φτάσουμε στο 25% τουλάχιστον. Εμείς πάντοτε είπαμε 30%. Ο δρόμος προς το Παρίσι πρέπει σε αυτόν να συμμετάσχουν όλοι, όλες οι χώρες. Από το 1990 έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος. Οι περισσότερες τώρα εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος περχόνται από χώρες που βρίσκονται στο κατόφλι της ανάπτυξης. Η Κίνα βλέπουμε ότι κινείται. Ελπίζω και η Ινδία και άλλες χώρες να ακολουθήσουν. Θα είναι μεν λιγότερα από ό,τι είχαμε ελπίσει στην Κοπενχάγη, δηλαδή η Παγκόσμια Συμφωνία με δεσμευτικούς στόχους. Τώρα ακούμε να μιλούν για nationally intended contributions, δηλαδή εθνικές συνεισφορές προθέσεων. Δηλαδή οι χώρες μέλη λένε τι επιθυμούν, τι προτίθεται να κάνουν, χωρίς όμως να αναλαμβάνουν υποχρέωση να το κάνουν. Πώς λοιπόν θα το στεγανοποιήσουμε, θα στεγανοποιήσουμε την προσπάθεια αυτή, ώστε να είναι δεσμευτικέ οι συμφωνίε αυτές για τελείως. Φοβούμαι ότι θα έχουμε ένα κείμενο με ωραία λόγια, αλλά το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο ωραίο. Πρέπει να ρωτήσω τώρα για τους πόρους που θα εισαχθούν στο Ταμείο του Πράσινου Κλίματος. Μου φαίνεται λίγο απίθανο να συγκεντρωθούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Μου φαίνεται απίθανο να μπορέσουν να το χρηματοδοτήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Υπάρχουν διάφοροι ειδικοί που εργάζονται πάνω σε διάφορα μοντέλα χρηματοδότησης, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες, ούτε κανεί ξέρει. Μήπως ο Γενικός Διευθυντής Ντεμπέκ γνωρίζει. Εκτός τώρα από τις κλασικέ προσπάθειες μετριασμού, mitigation δηλαδή, κάνουμε και άλλα πράγματα, όπω για παράδειγμα την αποδόμηση των επιδοτήσεων των ορυκτών ενεργειών. Το ίδιο για τους υδροχλωροφθοράνθρακες που και το ίδιο για το carbon pricing. Αυτά λοιπόν είναι πρόσθετα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν διότι αλλιώς δεν έχει προοπτικές επιτυχίες η συνολική προσπάθεια. Ευχαριστώ. Κύριε Γκερμπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Στελμπέκ για την καθαρή του σαφή του παρουσίαση. Προσέβλεπα στην διάσκεψη Μπανκιμούν στη Νέα Υόρκη, αλλά τώρα, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος στόχος του λέει ότι είναι οι παγκόσμιοι ηγέτες του κόσμου να επαναλάβουν τη δέσμευσή τους να έχουν αποτελέσματα το 2015 Όποτε επαναλαμβάνω κάτι που το έχουν ήδη υποσχεθεί, χαιρόμαστε εμένα, αλλά αυτό είναι το ότι παραπάνω, το περισσότερο που ελπίζουμε δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό. Επίσης δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτά που άκουσα, που έμαθα, ότι θα προσέλθουν λέει πάνω από 100 ηγέτες αλλά όχι πολλοί Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκών χωρών η κυρία Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός Κάμερον έχουν δηλώσει ήδη ότι δεν θα πάνε στη Νέα Υόρκη. Επομένως θα δώσουμε πολύ άσκημη εικόνα της ευρωπαϊκής Ηγεσία στα κλιματολογικά. Θα έρθει ο κύριος Μπαρόσο, αλλά όχι οι σημαντικότεροι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών μελών. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Ούστελμπέικ, τι σχεδιάζει να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό η Κομισιόν, θα πιέσει περισσότερο τους ηγέτες των χωρών της Ένωσης ώστε να προσέλθουν το Σεπτέμβριο στη διάσκεψη. Άλλα ερωτήματα. Περισσότερο για την εσωτερική ευρωπαϊκή διαδικασία. Είναι ατυχές βέβαια ότι δεν, έχουμε, δεν θα έχουμε κοινή ευρωπαϊκή θέση μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι θα δηλώσει ο κύριος Μπαρόσο λοιπόν ως ευρωπαϊκή θέση εκτός από το ότι δεν συμφωνούμε. και ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα ως πρωτοπορία για την αντιμετώπιση. Ποιο μήνυμα θα, μας, θα στείλει ο κύριος Μπαρόσο εκεί. Άλλο ερώτημα. Ποιες είναι οι προθέσεις της Κομισιόν για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Τι προτάσεις μπορούμε να αναμένουμε εκτός από τις προτάσεις για την περισσότερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τέλος για την ποιότητα των καυσίμων. Ευχαριστώ κύριο ότι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κευμπράντη. Όταν άκουσα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για το Σεπτέμβριο να μας μιλάει, φαίνεται ότι θα είναι μια συνάντηση οδυνηρή. Γιατί στα πλαίσια της διαδικασίας ε, της εντολής Μπαρόζο 1 ε, υπήρξε η στρατηγική του 2020 και στην Μπαρόζο 2 δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας. Αυτή θα είναι η τελευταία συνάντηση στην οποία ο Μπαρόζο θα μιλήσει για το κλίμα και δεν θα έχει κάτι να προσφέρει. Γι' αυτό θα είναι πολύ οδυνηρή η συνάντηση αυτή. Και για τον ίδιο τον ε, Μπαρόζο. Όταν ακούω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής θα απογοητεύομαι. Γιατί η φιλοδοξία μας θα είναι να επιβεβαιώσουμε κάτι το οποίο έχουμε ήδη επιβεβαιώσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Τι είναι αυτό το οποίο θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη. Τον Οκτώβριο θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Κορυφής, οπότε κανονικά θα πρέπει να πει κάτι για το 2030 και η Επιτροπή θα πρέπει και αυτή έτσι κι αλλιώς ε, να έχει κάτι να προσφέρει. Μια και θα φύγει ο Μπαρόσο τουλάχιστον να σπάρει μια φορά ένα ηγετικό ρόλο και ας πούν τις απόψεις τους. Και μια και δεν θα είναι και αρκετοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ο Μπαρόσο μπορεί να μιλήσει ελεύθερα και όχι να λέει λόγια κενά τα οποία, μας, τα οποία έχουμε συνηθίσει και τα οποία μόλις ακούσαμε και από εσά, κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής. Αν είναι να πει ο Μπαρόσο ότι έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα, στην ουσία τα ίδια ακούμε σαν μαγνητοφωνημένο μήνυμα εδώ και πολλά έτη, οπότε ίσως ε, αν είναι να πάει να πει αυτά, ας εξοικονομήσουμε το εισιτήριο και ας μείνει στις Βρυξέλλες ο Μπαρόσο. Αν πάει όμως θα πρέπει κάτι να πει, να πει κάτι πιο συγκεκριμένο, να μας πει τι θα κάνει για το 2030 θέματα τα οποία εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει στα λόγια, πρέπει να δώσει συγκεκριμένες υποσχέσεις. Θα πιέσει η Ευρώπη για διεθνή μέσα και όργανα έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις για το 2020 γιατί όλες οι συναντήσεις κορυφής στην ουσία επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία έχουν ήδη πει οι κυβερνήσεις με λίγα χρήματα, αλλά δεν υπάρχουν υποσχέσεις και επενδύσεις ε, για βελτιώσεις της κατάστασης μέσω πληρωμών σε τομείς όπως οι αερομεταφορές ε, και οι θαλάσσιες μεταφορές. Λοιπόν, ας μας μιλήσει τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο πολιετούς χρηματοδότησης και να μην περιμένουμε ε, κάθε φορά από το ΕΚΟΦΗΝ το τι θα γίνει του χρόνου. Λοιπόν, αν είναι να πάει ο Μπαρόσο να πει αυτά τα οποία έχει ήδη πει μέχρι τώρα, δεν χρειάζεται καθόλου. Ευχαριστώ. Τσουίκα. Hvala Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις ο κύριος Ντεμπέκερ, λέει η κυρία Σούισα. Είναι αλήθεια ότι η συνάντηση στο Παρίσι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την καταστροφή της Κοπενχάγης. Γι' αυτό είναι σημαντικές αυτές οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταθέσει τις θέσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς σαν Κοινοβούλιο. Να μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου είχε ε, θα έλεγα δεσμευθεί σε τρεις συγκεκριμένους στόχους. Ε, ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη οι στόχοι αλλά νομίζω ότι μέχρι το 2030 μπορούμε να ε, τους πετύχουμε για ε, το 2020 εξακολουθούμε να επιδιώκουμε την επιτυχία ορισμένων στόχων και είναι αλήθεια ότι η κατάσταση οικονομική αυξάνει τους κινδύνους και δεν λειτουργεί ο μηχανισμός ελέγχου όπως θα έπρεπε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί βοήθεια και προς τις ε, υποανάπτυξη χώρες. Έχει σημασία γιατί οι χώρες αυτές δεν έχουν τα απαιτούμενα μέσα και απαιτείται ο μηχανισμός για τη βοήθειά τους. Εμείς που είμαστε πιο αναπτυγμένοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος λοιπόν και θα πρέπει να προσέξουμε. Αναφέρομαι στις διεθνείς αερομεταφορές και στις εκπομπές επίσης των πλοίων είναι θέματα τα οποία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουμε. Πρέπει να προετοιμάσουμε λοιπόν σωστά τη συνάντηση κορυφής του Παρισιού έτσι ώστε να αποδειχθεί χρήσιμη. Λοιπόν, ε, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ζητούν το λόγο. Ο κύριος ακούγοντας τον κύριο Γενικό Διευθυντή, θυμούμε εκείνο το, το πνεύμα πρόθυμων εισάρξ ασθενής. Κάνουν προσπάθεια, έχουν πολλές ιδέες, αλλά όταν δω τι γίνεται για παράδειγμα για την αποδοτικότητα της ενέργειας, αυτά που είπε ο Πέτερ Λίζε, πρόκειται για πρόγραμμα συγκυρίας της βιομηχανίας και δημιουργεί απασχόληση και πρέπει να προωθήσουμε. Είναι καλό παράδειγμα. Ή επίσης η εμπορία των εκπομπών πρόκειται να αρχίσει λέει, το 2021, ενώ γνωρίζουμε ότι ήδη από το 2017 υπάρχει κίνδυνος να υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών στην αγορά. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσουν οι διεθνείς εταίροι στην περίπτωση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά ορισμένων χωρών μελών. Ελπίζω ο Μπαρόσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταφέρουν να συντονίσουν καλύτερα και για τη χρηματοδότηση. Είδαμε και στις τελευταίες διασκέψεις κορυφή του κλίματος Διάφορε χώρε μέλη να ανακοινώνουν διάφορα ποσά και να μην υπάρχει κανένα συντονισμός. Εγώ θέλω να υπάρξει καλύτερο συντονισμός για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τότε μπορεί να αποδώσει η προσπάθεια. Αλλιώ θα πάψουν να μας ακούνε καν στι διασκέψει κορυφή ούτε θα μα πιστεύουν, διότι βγαίνουμε και βγάζουμε κηρύγματα στις, στις ε, διεθνείς διασκέψεις, όμως μετά χωρίς να φταίει απόλυτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιστερούν οι χώρες μέλη, δεν, δεν έρονται στο ύψος των όσων έχουν ήδη δηλώσει. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λεπτομερή ενημέρωση που έκανε. ερώτηση. Πρώτα, για τους ευρωπαϊκούς στόχους για τις εκπομπές. Είναι σωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δίνει μόνο υποσχέσεις για την μείωση των εκπομπών. Πρέπει να λάβει πραγματικά μέτρα και να δείξει αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι πού βρίσκονται τα όρια των φιλοδοξιών αυτών. Εγώ άκουσα ότι το 2020 η μείωση των εκπομπών μπορεί να φτάσει και το 40%. Εδώ όμως μιλούμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για ένα συνολικό ποσοστό όλων των παγκόσμιων εκπομπών της τάξης του 13-14%. Όσο προσπάθεια και να κάνουμε εμείς δεν πρόκειται να βελτιωθεί η παγκόσμια εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ και Κίνα να αναλάβουν επίσης υποχρεώσεις και δεσμεύσεις συμφωνώ με τον Γενικό Διευθυντή ότι ένας στόχος θα πρέπει να είναι να πιστούν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ουσιώδη συνεισφορά και να πιέσουν Ενωμένες Πολιτείες και Κίνα να αναλάβουν και αυτές τις δεσμεύσεις. Δεύτερο, για την καθαρή ενέργεια. Εμείς που συμμετέχουμε εδώ στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος, νομίζω συμφωνούμε όλοι για την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων ενεργειών. Υπάρχουν όμως χώρες όπου η πυρηνική ενέργεια είναι καθοριστικός παράγοντας στο συνολικό μείγμα της ενέργειας. Για παράδειγμα στη Γαλλία ή και στη χώρα μου, την Ουγγαρία, που φτάνει και το 40% του energy mix. Υπάρχουν σχέδια να διατηρηθεί το ποσοστό αυτό συμμετοχή τη πυρηνική ενέργειας. Ερώτηση. Θεωρείτε ότι η διατήρηση ασφαλών πυρηνικών ικανοτήτων, safe nuclear capacities, είναι ένα θετικό βήμα προ την κατεύθυνση της ε, προστασία από την κλιματική αλλαγή. Έχει υπάρξει μια κάποια σύγχυση Ε, μιλάμε για το 40% της ε, αποδοτικότητας στην τομέα της χρήσης της ενέργειας και όχι των ανανεώσιμων πηγών. Λοιπόν, η κυρία Ράις έχει ζητήσει το λόγο. Α, η κυρία Ρίς τελικά ζητά συγγνώμη. Θα είμαι σύντομη, δεν θέλω να επιβαρύνω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με περισσότερες ερωτήσεις. Χαίρομαι που ξεκινάμε τις εργασίες μας με αυτή τη θεματολογία. Είναι μια θεματολογία στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος, αν και όπως ακούστηκε ε, αυτή η προσπάθεια έχει γίνει από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και όχι τόσο από το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει η συνάντηση κορυφής αυτή, η συνάντηση Μπαν στο τέλος του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντική και θα παίξει καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να καθοριστούν φιλόδοξες ε, προσδοκίες για το Παρίσι για να αποφύγουμε αυτά που συνέβησαν στην Κοπενχάγη αν και οι διαπραγματεύσεις όπως λέγουν ορισμένοι ξεκίνησαν ε, με λάθος τρόπο από ό,τι φαίνεται, ιδιαίτερα μέσω της πολωνικής κυβέρνησης η οποία δεν θέλει να παίξει με συλλογικό τρόπο το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει είμαι αρκετά αισιόδοξη. Πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα από ό,τι φαίνεται αλλάζουν γραμμή. Το είπε ο κύριος Ντεμπέκερ θα πρέπει ίσως να σταθούμε λίγο περισσότερο στο πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα. Και ένα τμήμα των εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματολογικές αλλαγές λέγουν ότι στην παρούσα φάση ότι έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο για να πετύχουμε τους στόχους του 2015 από ότι ήμασταν στην Κοπενχάγη και άκουσα και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας λέγει ότι ήδη είμαστε σε φάση ε, εκπλήρωσης των στόχων μείωσης ε, του, των εκπομπών διοξιδίου ε, σχετικά με τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που έχουμε για το 2020. Το θέμα είναι βέβαια και οικονομικό. Τι γίνεται με την χρηματοδότηση των μέσων που είναι απαραίτητα για να βοηθήσουμε τις χώρες του Νότου να αντιμετωπίσουν τις συνέχειες των κλιματολογικών αλλαγών. Και μία άλλη πιο πολιτική θα έλεγα και προοπτική ερώτηση. Άκουσα ότι ο κύριος Μπαρόσο θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνάντηση κορυφής. Ε, ε, σχετικά τώρα με τη Λίμα και το Παρίσι, διαρωτώ ε, τι μπορούμε να πούμε για την συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά έπαιξαν αρνητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και διαρωτώ με πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια κάποια συνεκτικότητα και μια κάποια ενότητα δράσης. Σα ζητώ συγγνώμη αλλά το όνομά σα το διάβασα στην αγγλική γλώσσα, χρειάζομαι χρόνο για να μάθω. Η κυρία Γκροστέτ έχει ζητήσει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειάζεται πολύ χρόνο για να συζητήσουμε τα κλιματολογικά και πολλές φορές έχουμε ξαναπεί τα ίδια με προηγούμενες συζητήσεις σε προηγούμενη θητεία. Ήταν μεγάλη απογοήτευσή μας στην Κοπενχάγη και η αποθάρρυνση που αισθανθήκαμε όλοι. Πρέπει όμως να παραμείνουμε ρεαλιστέ, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλυφθούν δεσμεύσει από τους εταίρους μας και πρέπει επίσης να αποφύγουμε να υπάρξει σύγχυση ως προς τα ποσοστά που αναφέρονται για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, για τις ανανεώσιμες, για τη μείωση των εκπομπών διότι ναι μεν δεσμευτήκαμε για 40% μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ενεργειακή αλλά πρέπει να επιμείνουμε και όλα. Για τα υπόλοιπα θα ήθελα να θυμίσω ότι η Ευρώπη ακόμη και αν είναι πρωτοπόρος σε αυτό το κλιματολογικό θέμα δεν είναι και τέλεια. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει έκθεση πρόσφατη που λέει ότι 70% των εκπομπών στον κόσμο προέρχεται από ηλεκτρικούς σταθμούς που κινούνται με άνθρακα. Και στην Ευρώπη υπάρχουν από τις πιο μολυντικές τέτοιες μονάδες, στην Πολωνία, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Πρέπει και εκεί να κάνουμε μια προσπάθεια, ώστε η σταθμή αυτή, φυσικά δεν ζητάω να απαγορευτεί η χρήση του άνθρακος γιατί το κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να αποφασίσει μόνο του ποιες ενεργειακές πηγές θα χρησιμοποιήσει, αλλά να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τεχνολογία καθαρότερη. Γνωστά τα παραδείγματα, τα εξετάσαμε πριν από 6 χρόνια, το 8 και θα ήθελα να γνωρίζω πού βρισκόμαστε, τι τεχνολογία χρησιμοποιείτε, πώς αποθηκεύεται και αν αποθηκεύεται το διοξίδιο. Έχει προχωρήσει καθόλου αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε επίσης αν θέλουμε να εισακουστούμε από τους εταίρους μας να δείξουμε ότι και εμείς προχωρούμε στη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει και η έρευνα για την αποθήκευση της ενέργειας. Πώς οι ενεργειώσιμες πηγές θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικές γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι και πολύ αποτελεσματικές, επιχορηγούνται και παρόλα αυτά δεν είναι αποτελεσματικές γιατί δεν μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε. Αν βρεθεί κάποια τέτοια νέα τεχνολογία πρέπει να την γνωστοποιήσουμε και στους εταίρους μας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πού βρισκόμαστε για τις τεχνολογίες αυτές, αν προχωράμε ή όχι. Επίσης μερικά στοιχεία για την ε, εκμετάλλευση του λεγόμενου πράσινου ταμείου που θα ζητηθεί στη Λίμα όπως είπατε, αλλά θέλω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες ερωτήσεις έχω προς τον κύριο Ντεμπέκε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2007 τα Ενωμένα Έθνη εξέδωσαν έκθεση που λεγόταν The Long Shadow of Livestock με συμμετοχή του καθηγητού Φένικ στην έκθεση αυτή είχε αποδειχθεί ότι πάνω από 18% των εκπομπών που είναι βλαβερές για το κλίμα προέρχονται από την παγκόσμια κτηνοτροφία. Κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και στις ε, διασκέψεις κορυφής των Ενωμένων Εθνών αλλά και στην προπαρασκευαστική διάσκεψη για τη Λίμα αλλά και για το Παρίσι στο σημαντικό αυτό τομέα που είναι όπως είπα σημαντικό για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στο πολύ σε δύο βαθμούς. Πεντιτσίνη ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω αυτά τα οποία είπε ο παρακαθήμενος μου. Φυσικά και θα συμφωνήσω για τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει στον τομέα της αποδοτικότητας της ενέργειας, αλλά πράγματι υπάρχει μια αντιφατική στάση από ορισμένα κράτη, τα οποία επιμένουν να χρησιμοποιούν ενέργειες, ε, ε, μορφές ενέργειας που δεν είναι αυτές οι οποίες καθιστούν πιο αποδοτική την παραγωγή της ενέργειας. Η Ιταλία σαν παράδειγμα η οποία περιέργως ε, και μέχρι το 20 θα βασίζεται στο πετρέλαιο, σε ορυκτά καύσιμα. Στόχος της Ιταλίας για το 2020 είναι να διπλασιάσει την παραγωγή ε, ε, πετρελαίου και στην υπηρετική χώρα και σε θαλάσσιες περιοχές. Και μάλιστα και με τεχνικές και μεθόδους ε, οι οποίες ε, πλέον έχουν ξεπεραστεί και απαγορεύονται στον υπόλοιπο κόσμο όπως το λεγόμενο fracking. Συνεπώς λοιπόν όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα του τουρισμού γιατί αυτή η αναζήτηση θα γίνει στην ε, Σικελία, στην Καλαβρία, στην Απουλία και στην Αδριατική θάλασσα, τουριστικές περιοχές. Το θέμα είναι να δούμε λοιπόν πώς θα ξεπεράσουμε αυτές τις αντιφάσεις των κρατών μελών, μιας και οι στόχοι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ιδιαίτερα υψηλοί. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος. Κλείσαμε λοιπόν με τον κατάλογο των ομιλητών. Νομίζω ότι συνολικά αυτό το οποίο βγαίνει από τις παρουσιάσεις των συναδέλφων είναι μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με πιο ισχυρό τρόπο. Από την άλλη έχουν κατατεθεί και συγκεκριμένα ερωτηματικά και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον Διευθυντή της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κυριότερο ερώτημα ήταν τι θα πει ο Πρόεδρος στη διάσκεψη Μπαν Κιμούν. Αλλά δεν το ξέρω, δεν μπορώ να μαντέψω τι προτίθεται να πει. Φαντάζομαι θα πει ότι η Ένωση έχει ήδη μακρά παράδοση για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Στο Κιώτο έχει αναλυφθεί η δέσμευση να τα μειώσει κατά 8% μέχρι το 12% η Ένωση μείωσε τις εκπομπές της κατά 18%. 18%. Μετά από αυτή την πρώτη περίοδο άρχισε η δεύτερη. Και τώρα συμπληρώνουμε τους στόχους για το 2030, δηλαδή 40% μείωση, 20% παραπάνω από ό,τι οι στόχοι του 20. 27-28, τουλάχιστον 27% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Δεν ξέρω τι θα πούν οι νέοι επίτροποι, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι υψηλότερα από το 25%. Πιστεύω ότι η Ένωση έχει μακρά παράδοση λοιπόν στη μείωση των εκπομπών και αποτελεσματικότητα. οι επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου αναμονάδα ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά το μισό. Και γι' αυτόν τον λόγο η Ένωση συνομιλεί με άλλες μεμονωμένες χώρες όχι μόνο για συνεννόηση γενικότερα αλλά και για να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της ως παράδειγμα. Στην Κίνα ας πούμε υπάρχουν 7 πιλωτικά προγράμματα για την εμπορία των εκπομπών που τη, πρόγραμμα που το στήριξαν οι Ευρωπαίοι και οι Κομισιόν και πολλές ιδέες και λογισμικά έχουν χορηγηθεί στους Κινέζους. Σήμερα λοιπόν στο Σέντζεν οι τιμές στην αγορά είναι διπλάσιες από την Ευρώπη και αυτό δείχνει ότι και άλλοι στον κόσμο ακολουθούν την οδό που χαράξαμε εμείς. Οι τιμές στην αγορά άνθρακα είναι χαμηλές, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχει μία πρόταση σχετικώς και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας σύντομα να δεχτούν αυτή την πρόταση. Όσο για τα βασικά μέτρα που λάβαμε στην Ένωση όπως το ETS, μας μιμούνται πολύ και στην Κορέα και στην Καλιφόρνια και στις Ηνωμένε Πολιτείε και αλλού για την εμπορία των κομπών δηλαδή. Στην Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ προετοιμάζεται νομοσχέδιο αφού έγινε προσφυγή για το κατά πόσον είχε το δικαίωμα να το πράξει. <clears throat> Αυτό λύθηκε όμως τώρα. Προετοιμάζει λοιπόν προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ιδιαίτερα από καύση άνθρακα από σταθμούς ηλεκτρο... παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΙΠΑ υποσχέθηκαν λοιπόν 17% μείωση στην Κοπενχάγη και σχεδόν το έχει πετύχει αυτή τη στιγμή, όπως και εμείς το στόχο μας του 20% για το 2020. Το σημαντικό ερώτημα λοιπόν που επίσης θα θέσει ο κύριος Μπαρόσο νομίζω είναι ότι είναι σημαντικό περισσότερες χώρες στον κόσμο να ζητήσουν περισσότερη μείωση, να έχουν πιο φιλόδοξους στόχους. Όχι μόνο λόγω της επιτυχίας των δικών μας μέτρων, το μερίδιο των εκπομπών <clears throat> διοξιδίου <clears throat> διεθνώς από το 13% έχει φτάσει στο κάτω από το 10% θα φτάσει μέχρι το 2030. Αυτά βέβαια δεν θα πετύχουν παρά μόνο αν και άλλοι ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο οι νέες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία των Παρισίων πρέπει να έχουν ως βάση τη λέξη και την έννοια της συμμετοχής. Περισσότερες χώρες πρέπει να συμμετάσχουν στα προγράμματα μείωσης των εκπομπών και αυτό μπορεί να απαιτήσει και ορισμένες υποχωρήσεις για τι πράγμα θα δεσμευτούμε στο Παρίσι. Μήπως είναι επαναχώρηση σχετικά με αυτά που είπαμε στο Κιώτο. Ίσως να είναι κάποια επαναχώρηση σε σύγκριση με το Κιώτο, αλλά προσπαθούμε πάρα πολύ η κύρια πρόταση των Παρισίων να είναι μια σημαντική μείωση των εκπομπών και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων να συμπεριλαμβάνουν και επιτήρηση και εποπτεία της εφαρμογής των δεσμεύσεων με μεγάλη διαφάνεια ώστε όλοι να μπορούμε, όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να ελέγχουν τι συμβαίνει. Αυτό το MRV, Monitoring Reporting and Verification, θα είναι το, στο κέντρο των συζητήσεων στο Παρίσι. Και όπως λένε όλοι θα είναι από τα κυριότερα στοιχεία και του τελικού κειμένου της Λίμας. Με βάση λοιπόν τα πεπραγμένα μας γνωρίζοντας ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα στόχο δηλαδή 40% θέλουμε να υπάρχει ένα σύστημα μεγάλης διαφάνειας με βάση το MRV που σας έλεγα. Πολλά ερωτήματα αφορούσαν τη χρηματοδότηση των μέτρων κλιματολογικής αντιμετώπισης. Σε τι βαθμό δηλαδή στο πράσινο κλιματολογικό ταμείο υπήρξε πρόοδος. Μπορεί να αρχίσει ήδη η κεφαλαιοποίηση του. Έχουν αρχίσει ήδη τα πρώτα μέτρα και θα γίνει σε λίγο απέτηση της Συμφωνίας των Παρισίων. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι το κατά πόσον η χρηματοδότηση που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει για την κλιματολογική αντιμετώπιση έχει οδηγήσει σε πραγματική μείωση των εκπομπών. Στα πλαίσια των συζητήσεων του Ταμείου αυτού έγινε λόγος και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας. Όλες οι χρηματοδοτήσεις έχει εξεταστεί αν έχουν δαπανηθεί σωστά και αν υπήρχαν αποτελέσματα. Αυτό το κάναμε και με τα χρήματα που δαπανά η Κομισιόν για την αναπτυξιακή συνεργασία που έχει σαν πολύ σημαντικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα. Το ίδιο γίνεται και με την λεγόμενη κλιματολογική συμμαχία. Όλα αυτά βασίζονται σε ελέγχους για την αποτελεσματικότητα. Αν πράγματι γίνεται ό,τι υποτίθεται ότι θα γινόταν. Επίσης υπήρξε ένα ερώτημα για το energy mix που χρησιμοποιούν οι διάφορες χώρες. Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας, του άνθρακα, του πετρελαίου και του αερίου καθώς και του σχιστολιθικού αερίου. Αυτό είναι θέμα των χωρών μελών. Δεν είναι δουλειά της Κομισιόν να επιβάλλει ή να δηλώσει τι πρέπει να κάνουν οι χώρες μέλη. Αυτό είναι εθνική δικαιοδοσία. και πολλά χρόνια έτσι θα είναι ακόμα. Τι θα μπορούσαν να κάνουν όμως είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων του 2030, δηλαδή να υπάρξει ένα σύστημα διακυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα. Χρειάζεται πολύ περισσότερη διαφάνεια για τα σχέδια των χωρών μελών και προς τους γείτονές τους. Και αυτό θα είναι μεγάλο όφελος για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για την κλιματολογική πολιτική, αλλά και για την ενεργειακή. οι αποφάσεις για την πυρηνική ενέργεια που θα εφαρμοστούν σύντομα στην Ευρώπη θα σημάνουν κάποια μείωση σχετική, αλλά η χρήση του άνθρακα λυπούμαστε γιατί έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, διότι ο άνθραξ είναι φτηνός και ελπίζουμε και αυτό να το αντιμετωπίσουμε μέσω καλύτερης λειτουργίας της αγοράς του άνθρακα. Επίσης τέθηκε ένα ερώτημα για την αποθήκευση των διοξιδίου. Μερικές χώρες μέλη το πειραματίζονται ήδη. Η Κομισιόν μόλις αποφάσισε μέχρι 300 εκατομμύρια ευρώ να δοθούν για ένα πρόγραμμα αποθήκευσης του διοξιδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρξε, τέθηκε και ένα θέμα για τη γεωργία. Αυτό είναι τμήμα διεθνών διαπραγματεύσεων που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει. Θέλουμε περισσότερη συλλογή πληροφόρησης και συζητούμε το θέμα αυτό με τους συναδέλφους μας που ασχολούνται με την κοινή αγροτική πολιτική καθώς και με τον πυλώνα 2 για να δούμε κατά πόσον οι αγροτικές πρακτικές χρησιμοποιούν λιγότερο εκπομπές διοξιδίου. Είχαμε πει για τη δήλωσή μας, την ανακοίνωσή μας για το 2030 ότι θα θέλαμε ίσως να συνδυάσουμε τις εκπομπές από τη γεωργία και τη δασοκομεία χωριστά από εκείνες που διαπιστώνονται για την ενέργεια. Άλλο ερώτημα αφορούσε τις διαρροές διοξιδίου. Carbon leakage δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ανακοίνωση που έλεγε ότι θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον κατάλογο τομέων όπου διαπιστώνεται διαρροή μέχρι το 2020. Αυτό θα έπρεπε να καθησυχάσει όσους ανησυχούν στη βιομηχανία γιατί πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της διαρροής μετά το 2020. Η αξιολόγηση του δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό σήμερα, αλλά εν ώψη του 2030 και ανάλογα με το αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων δεν το ξεχνάμε και οι ηγέτες επιχειρηματίες και βιομήχανοι ούτε εκείνοι το ξεχνάνε. Υπάρχει λοιπόν συζήτηση για τη διαρροή και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και σήμερα στους τομείς που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο όπου διαπιστώνεται διαρροή χορηγούμε περίπου τα μισά ποσά που υπάρχουν για την αγορά του άνθρακα. Επίσης ερώτημα υπήρξε για την επικύρωση του KP2 της δεύτερης περίοδου του Κιώτο δηλαδή. 27 χώρες μέλη συμφώνησαν να προχωρήσουμε αλλά περιμένουμε ακόμη να το συμφωνήσουν όλες και οι 28 η δηλαδή. Ελπίζουμε τον Οκτώβριο να υπάρξει συμφωνία και γι' αυτό. Επίσης ερώτημα γιατί προτάσεις συζητιούνται ή προετοιμάζονται από την Κομισιόν. Αυτό που προετοιμάζεται είναι το απόθεμα σταθερότητας της αγοράς του άνθρακα. Επίσης υπάρχει πρόταση για την μέτρηση των εκπομπών από τον τομέα των θαλασσίων δραστηριοτήτων και μεταφορών και λεπτομέρειες για τη δέσμη του 2030 αλλά περιμένουμε γι' αυτό τον Οκτώβριο τις αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων διότι ανάλογα με αυτό θα προετοιμάσει η Κομισιόν την ομοθεσία της για την αγορά του άνθρακα και του διοξιδίου του άνθρακα και αν χρειαστεί να αλλάξει τίποτα πέρα από την πρόταση για τη σταθερότητα της αγοράς θα γίνει. Ίσως να συζητηθούν και πανενοσιακά μέτρα για τη διευκόλυνση της μείωσης των εκπομπών σε σχέση με τα αυτοκίνητα, με τα καύσιμα με τα βιοκαύσιμα και γενικά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να καταλήγουν σε εκπομπές όπως παραδείγματο χάρη τα air conditioning που μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα. Νομίζω ότι με αυτά απάντησα στα περισσότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί, ίσως όχι με αρκετή λεπτομέρεια, αλλά θα ήθελα να σας ε, ησυχάσω ότι στην διάσκεψη Μπάνκιμον έχουμε τι να πούμε, έχουμε τα πεπραγμένα μας και την αποτελεσματικότητά μας και αυτό θα αποδείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στο δρόμο που χαράξαμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Ντεμπέκερ, τον διευθυντή Ντεμπέκερ. Νομίζω ότι με τις απαντήσεις τις οποίες μας δώσατε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει κλείσει πλέον το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω εδώ μαζί μας τον συνάδελφο κύριο Νίκολσον, ο οποίος είναι ο εισηγητής για το επόμενο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, τα νέα τρόφιμα. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε χωρίς καθυστέρηση να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Όπως γνωρίζετε όλοι, η νομοθετική ε, διαδικασία για τα novel foods έχει μια μακρά ιστορία. Το 2008 υιοθέτησε την πρώτη πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κανονισμός δηλαδή, αλλά κατά τη διάρκεια της κανονικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Και στο τέλος των εργασιών τον Μάρτιο δηλαδή της ε, ομάδας ε, διαπραγμάτευσης δεν είχαμε μια αποδεκτή πρόταση από πλευράς του Ευρωπαίου νομοθέτη και έτσι έκλεισε η διαδικασία. Κάποια θέματα όμως παρέμειναν σε... έμειναν ανοιχτά ε, συγκρούσεις αρμοδιοτήτων όπως θυμάται ο προκατοχός μου πάρα πολύ καλά για την κλωνοποίηση είχαμε πολλά προβλήματα ε, για το ποιος έχει την κύρια αρμοδιότητα με την Επιτροπή Γεωργίας. Και τώρα ε, έχουμε επανέλθει στη νέα πρόταση η οποία διατυπώθηκε αυτή τη φορά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσω ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου ε, ζητήθηκε να υπάρξει μια μελέτη επιπτώσεων και οι εργασίες μας αυτό θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να δώσουμε πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει την πρότασή της για τα νέα καινοτόμα τρόφιμα. Μετά θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της ΕΦΣΑ και όλων των, όλους τους εμπειρογνώμονες που έχουν συντάξει την έκθεση και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση στο εσωτερικό της Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο ξεκινώντας στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει την πρότασή της. Η κυρία Σαντάλ Μπρούση. Έχετε το λόγο. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Σαντάλ Μπρούτσι. Πάντως είχα καταλάβει ότι ε, εμένα εννοούσατε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ επίσης που βάλατε το σημαντικό θέμα στην ημερησία σας διάταξη σήμερα. Ευχαριστώ και στον εισηγητή κύριο Νίκολσον Είπατε σωστά ότι η συνδιαλλαγή απέτυχε και ιδίω για θέματα που σχετίζονται με την κλωνοποίηση έχουμε συντάξει αυτή την πρόταση για τα νέα τρόφιμα και υπάρχουν και δύο προτάσεις βέβαια για την κλωνοποίηση. Είναι σημαντικό να συζητηθεί η πρόταση διότι αυτή διαλαμβάνει τα περισσότερα από τα θετικά αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής και ο κανονισμός περί νέων τροφίμων, novel food, όσο έχει σήμερα, αναφέρεται σε νέα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν καταναλωθεί σημαντικά στην Ευρώπη. Επίσης, τρόφιμα τα οποία οι επιχειρήσεις θέλουν να διαθέσουν στις αγορές. Άρα, ο κανονισμός έχει ως στόχο την διευκόλυνση της διάθεση στην αγορά αυτών των novel food, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι ασφαλή και ε, ενισχύοντας και την καινοτομία και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο κανονισμός που ισχύει σήμερα από στα μάτια πολλών και της βιομηχανίας και των καταναλωτών αλλά και ημών των policy makers δεν είναι αποτελεσματικός. Είναι μακρές οι διαδικασίες, η έγκριση περνάει πρώτα από τις χώρες μέλη, αν αυτές έχουν ενστάσεις τότε διαβιβάζονται οι φάκελοι μεταξύ των χωρών μελών. Μετά στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν χρειάζεται ιδιαίτερη επιστημονική μελέτη πηγαίνει στον οργανισμό ΕΦΣΑ. Δηλαδή διαδικασία χρονοβόρος και όλοι θεωρούν ότι μπορεί να βελτιωθεί. Γι' αυτό και καταθέσαμε την πρόταση αυτή, όπως είπατε και εσείς, απέτυχε στην ε, συνδιαλλαγή και τώρα έχουμε κατέβει με νέα πρόταση. Για να υποστηρίξουμε την καινοτομία κάνουμε καλύτερες τις διαδικασίες, δηλαδή οι αιτήσει διαβάζονται πλέον ευθέως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται ε, η αξιολόγηση του κινδύνου από την ίδια την ΕΦΣΑ για να αποφευθούν οι μακρές οδοί που σας ανέφερα προηγουμένως. Άρα θα κινείται ταχύτερα η διαδικασία και θα διευκολύνει σημαντικά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Δηλαδή αγροτικών προϊόντων που δεν έχουν καταναλωθεί ποτέ στην Ευρώπη ως τώρα επειδή όμως είναι αγροτικά προϊόντα και εάν για παράδειγμα έχουν καταναλωθεί σε αυτή την τρίτη χώρα επί μια 25 ετία προτείνουμε στην τρίτη χώρα και κυρίως αυτές είναι αναπτυσσόμενες χώρες να μην περάσουν μέσα από την διαδικασία έγκρισης ή αδειοδότησης αλλά από μια διαδικασία κοινοποίηση, διαδικασία πιο light και πιο γρήγορη. Βέβαια οι χώρες μέλη πάντα θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν ενστάσεις εάν υπάρχουν σοβαρά θέματα ασφάλειας. Και τότε βέβαια το προϊόν καταλήγει στην ΕΦΣΑ. Για να δοθεί όμως η δυνατότητα αυτή στις τρίτες χώρες για αγροτικά προϊόντα τα οποία οι ίδιες έχουν καταναλώσει επί ένα διάστημα, περιλαμβάνεται αυτό το καινοτόμο στοιχείο στην πρόταση. Ο ορισμός του novel food είναι επίσης ένα νέο καινοτόμο στοιχείο. Θελήσαμε να απλουστεύσουμε τον ορισμό είναι επομένως νέο τρόφιμο, novel food, δεν έχει καταναλωθεί ποτέ στην Ευρώπη από το 1997, δεν έχει καταναλωθεί ούτε σε σημαντικό βαθμό σε κάποια χώρα μέλος και θέλουμε να αποφύγουμε τη δυσκολία ταξινόμησης των novel food. Έχουμε λοιπόν ένα διοικητικό κατάλογο αυτών των νέων τροφίμων που εμπίπτουν στον ορισμό. Βέβαια εδώ μπορεί να προκύψει κάποια σύγχυση. Δεν υπάρχει δηλαδή πλήρης ξεκάθαρος κατάλογος των ε, νέων τροφίμων, αλλά υπάρχει περισσότερο μια απεικόνηση και θέλουμε γι' αυτό να ε, αποφύγουμε την, την ε, σύγχυση αυτή. Για την ίδια διαδικασία τώρα είναι σημαντικό να σημειώσει κανείς ότι η αδειοδότηση μέσα στην πρόταση θα είναι γενικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ιδίω οι μικρέ και μεσές επιχειρήσεις δεν θα έχουν τόσο εύκολα τα μέσα να προχωρήσουν, να ζητήσουν πλήρες risk assessment. Υπό την ισχύ του παρόντος κανονισμού υπάρχει και μια διαδικασία που επιτρέπει σε άλλες επιχειρήσεις να μπουν σε μια αγορά για ένα εγκεκριμένο σύστημα αλλά αυτή τη στιγμή έχει αδειοδοτηθεί ένα novel food υπό την ισχύ του παρόντος κανονισμού ή συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν που θέλει να διαδίδει στην αγορά είναι παρόμοιο, είναι ισότιμο με το ήδη αδειοδοτημένο προϊόν. Για την διαδικασία την ίδια ίσως έχετε σημειώσει ότι προβλέπουμε προθεσμία πέντε μηνών για την ΕΦΣΑ για... και επίσης έχουμε προθεσμία 9 μηνών για την αδειοδότηση. Για την προστασία δεδομένων τώρα υπάρχει πάλι μια γενική αδειοδότηση όπως είπα, αλλά για να ενισχύσουμε ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την ικανότητα ή μπορούν να επινοήσουν στη βάση, να φεύγουν δηλαδή στην βάση των ερευνών τους νέα τρόφιμα, τους προτείνουμε μια προστασία. Δεν θα είναι δηλαδή γενική αδειοδότηση, θα είναι η επιχείρηση εκείνη που θα μπορεί να προσφέρει το τρόφιμο στην αγορά γιατί έχει κάνει την ίδια, ίδια την έρευνα. Πρέπει όμως η ίδια να είναι η διοκτήτρια των δεδομένων. Να, γνωρίζει, δηλαδή, να μπορεί να αποδείξει δηλαδή ότι αυτή ε, διαθέτει τα σχετικά δεδομένα. Όπως είπα, Αυτό επιτεύχθη ε, ως αρθετικό αποτέλεσμα από τη συνδιαλλαγή και είπατε κι εσείς βέβαια ότι εκεί το μέγα εμπόδιο, εμπόδιο ήταν η κλωνοποίηση. Θα βελτιώσουμε το υφιστάμενο σύστημα γιατί όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται βελτίωση. Θέλουμε να το επιταχύνουμε επίσης για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά καθώς επίσης και την καινοτομία διατηρώντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των τροφίμων. Λάβαμε χθε και ευχαριστούμε την γραμματεία του Κοινοβουλίου λάβαμε το σχέδιο μελέτης αντικτύπου, το οποίο διαβάσαμε. Θα περιοριστώ σε αυτά για την ώρα και ευχαρίστως θα απαντήσω σε ερωτήσεις εφόσον έχετε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάντως που εγγράψατε το θέμα στην ημερησία σας διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας καλέσατε σε αυτή την συζήτηση. Η ΕΦΣΑ καταρχάς δεν ε, δημιουργεί νομοθεσία, ούτε είναι υπεύθυνη για την χάραξη πολιτικής. Θα ήθελα να τονίσω μερικές από τις δραστηριότητες της, τωρινές και μελούμενες, για την, ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας που εσείς αποφασίζετε. Στην αποκεντρωμένη διαδικασία η ΕΦΣΑ αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος έχει εκφράσει διαμαρτυρία ή παράπονο, ένα τρίτο δηλαδή των αιτημάτων ή των αιτήσεων που έχουν αξιολογηθεί από την ΕΦΣΑ και αυτό δείχνει ότι η νέα πρόταση με την αποκεντρωμένη διαδικασία θα επιταχύνει τα πράγματα για την αξιολόγηση των προτινομένων novel funds. Επίσης θέλω να τονίσω ότι η υπηρεσία αυτή χορηγείται δωρεάν από την ΕΦΣΑ. και για τα novel funds εκτιμούμε ιδιαίτερα το ότι η διαδικασία αυτή η αποκεντρωμένη θα επιταχύνει τα πράγματα, από την άλλη όμως θα αυξήσει και το άχθος εργασίας στον μόχθο της ΕΦΣΑ. Θα ανακατανύμουμε το προσωπικό μας και αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να ζητήσουμε νέες προσλήψεις. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι μετά το αίτημα της Κομισιόν αρχίσαμε να προετοιμάζουμε τα έγγραφα, των οδηγό για την υποβολή αιτήσεων από τις χώρες μέλη και θα έχει τυπωθεί και διανεμηθεί τον Οκτώβριο. Εφόσον βέβαια εγκριθεί η νέα νομοθεσία για τα Novel Funds. Θα γίνει και δημόσια διαβούλευση ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να αποφανηθούν και τα σχόλια αυτά θα συμπεριληφθούν, θα ληφθούν υπόψη στα τελικά οδηγητικά κείμενα. Οι ετούντες και χώρες μέλη, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, μέχρι το 16 θα τύχει πληροφόρησης για να υπάρξει μεγαλύτερη αποσαφήνιση των κειμένων των καθοδηγητικών κειμένων και για να γνωρίζουν οι ετούντες ποιες ακριβώς είναι οι επιστημονικές απαιτήσει για να κάνει κανείς μια αίτηση για Novel Fund. Επίσης η ΕΦΣΑ πρόσφατα, σύμφωνα και με την πρόσφατη νομοθεσία, θεωρεί ότι στο μέλλον μπορεί ο ετών να ζητάει περισσότερες πληροφορίες και κατά τη διάρκεια της αποτίμησης του προϊόντος του. Γνωρίζουμε ότι πολλές χώρες μέλη έχουν εμπειρία επιστημονική για την αποτίμηση θεμάτων Novel Fund και θεωρούμε ότι καλό θα ήταν την εμπειρία τους αυτή να τη συνεχίσουν, να, παίζουν, να συνεχίσουν να παίζουν δηλαδή συμβουλευτικό ρόλο για τους ετούντες εφόσον βέβαια έχουν την τεχνογνωσία για να κάνουν την πρώτη ιδιωτική τους μεμονωμένη αποτίμηση. Εμείς σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα είδος συμβολέου όταν θα εγκριθεί η νομοθεσία και οι χώρες μέλη να υποστηρίξουν την ΕΦΣΑ για τις προπαρασκευαστικές έρευνες, πράγμα που θα μας βοηθήσει και θα επιταχύνει πολύ τη δουλειά μας. Επίσης, στο συμβουλευτικό βήμα τον περασμένο μήνα, συζητήσαμε τα γενικά θέματα και προβλήματα που μπορούμε να συνδυάσουμε με τους εμπειρογνώμονες των χωρών μελών αλλά όπως γίνεται συχνά στην ΕΦΣΑ είναι και ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ΕΦΣΑ για την παρουσίασή της. Τώρα ο εκπρόσωπος του Κέντρου για τη Στρατηγική είναι το κέντρο που με τους Τόμσινγκ, Ρίτσαρτον και Μάλλατ είναι αυτοί οι οποίοι ε, συνέταξαν μία μελέτη την οποία θα μας παρουσιάσουν. Έχετε 15 λεπτά, μπορείτε να τα διαχειριστείτε μεταξύ σας. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε εδώ σήμερα για τη μελέτη αυτή των επιπτώσεων. Έχουμε επίσης και τον συνάδελφο Τόνκιν από την ΕΙΝΤΑΣ του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα σας δείξουμε ποιες είναι οι βασικές, τα βασικά ευρήματα της μελέτης την οποία κάναμε. Θα ήθελα κάποιος να ξεκινήσει τις διαφάνειες. Μας δόθηκε λοιπόν μια εντολή η οποία είχε τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον να αναθεωρήσουμε ε, την μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008. Δεύτερον να εξετάσουμε την πρόταση η οποία βρίσκεται υπό εξέταση, τα ωφέλη, και δεύτερον να δούμε τι νέο υλικό έχει δημοσιευθεί πρόσφατα από το 2008 και μετά που είχε γίνει προηγούμενη μελέτη. Κάναμε αρκετές ερευνητικές ε, δράσεις ε, και σε επίπεδο εξέτασης της φιλολογίας που υπάρχει γύρω από τα θέματα αυτά και κάναμε και ένα πρόγραμμα με συνεντεύξεις που κάλυψε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κοινοτικά σώματα, την ΕΦΣΑ, τις αρμόδιες ε, αρχές στα διάφορα κράτη-μέλη, ενώσεις παραγωγών, ενώσεις καταναλωτών κτλ. Φυσικά ήρθαμε σε επαφή όπως είπα και με εκπροσώπους των καταναλωτών και άλλους εμπλεκομένους. Πάρα πολύ σύντομα τώρα τα κεντρικά θέματα στα οποία σταθήκαμε δεν θα τα αναλύσω με λεπτομέρεια. Οι συνάδελφοι θα ασχοληθούν με τα θέματα αυτά λεπτομερέστερα. Υπήρξαν όμως πέντε βασικά θέματα που αφορούσαν την εμβέλεια και τον ορισμό της έρευνας αυτής, διαδικασίες ε, επικεντρωμένες αδειοδότησης, αποτελεσματικότητα του συγκεντρωτικού συστήματος, ο ρόλος των εθνικών αρχών και οι σχέσεις με άλλες απαιτήσει διακανονιστικού τύπου. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να πω ότι παρουσιάσαμε μία πρόταση έκθεσης η οποία είναι διαθέσιμη και η οποία θα πάρει την τελική της μορφή σύντομα μετά από την παρουσίαση εδώ και είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμκινς τώρα, ο οποίος θα ασχοληθεί με τα υπόλοιπα θέματα. Η επόμενη διαφάνεια, λέει ο κύριος Τόμκινς, στόχος και ορισμοί, εμβέλεια και διορισμοί. Ήδη ξεκινήσαμε από την πρώτη οδηγία του 97 διαμορφώσαμε τις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες ε, μας επιτρέπουν να λάβουμε υπόψη τα νέα προϊόντα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον στην αγορά. Όταν ήρθαμε σε επαφή με τους καταναλωτές είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πολλοί πιστεύουν ότι οι νέοι ορισμοί θεωρούν ότι πάρα πολλά προϊόντα, χιλιάδες προϊόντα πρέπει να τύχουν μια νέα μορφή διοδότησης πλέον. Ιδιαίτερα τα προϊόντα τα οποία κυκλοφόρησαν πριν από το 15 ε, Μαΐου του 2097 είχαν θεωρηθεί νέα προϊόντα όπως ε, νέες ποικιλίε ε, φρούτων όπως επίσης και διασταυρούμενες ποικιλίε πρέπει να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό βάρος όταν ζητούν αδειοδότηση ή παραγωγή και υπάρχει μια νομική αβεβαιότητα. Οι καταναλωτές έχουν μια άλλη άποψη. Θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες παράνομες δυνατότητες εισαγωγής αυτών των προϊόντων χωρίς αδειοδότηση. Υπάρχουν λοιπόν απόψεις οι οποίες διήστανται μεταξύ τους και βασικός μας στόχος εδώ, βασική μας σύσταση μάλλον, είναι να υπάρξει περισσότερος διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τους καταναλωτές, τις οργανώσεις των καταναλωτών, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς επιπτώσεις ε, ε, δημιουργούν οι νέοι αυτοί ορισμοί. Οι επιπτώσεις λοιπόν στην διαδικασία κεντρικής αδειοδότησης ε, είναι οι εξής. Ε, η αρχική ε, γνωμοδότηση θα προέρχεται από την ΕΦΣΑ. Θα συγκεντρώνουμε και τις αξιολογήσεις τις οποίες κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χάνουμε πάρα πολύ χρόνο όταν ζητείται η κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ενώ στο παρελθόν υπήρχαν απαιτήσει για χιλιάδες που λέει ο λόγος επιστημονικές απόψεις, τώρα απαιτούνται πολύ λιγότερες. Η διαδικασία επιτροπολογίας βέβαια παραμένει να είναι πάρα πολύ αργή και μπορεί στις μόνιμες επιτροπές να υπάρξουν καθυστερήσεις. Γι' αυτό λοιπόν εάν πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σοβαρή σε σχέση με την αξιοπιστία της διαδικασίας θα πρέπει να σεβαστεί ένα αυστηρόχρονο διάγραμμα συγκεκριμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακούσαμε επίσης και για τις νέες απλοποιημένες διαδικασίες και για τα παραδοσιακά προϊόντα όταν υπάρχει ένα προϊόν από άλλη χώρα το οποίο θεωρείται ασφαλές και το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς ε, ε, καταναλωτές, τότε μπορεί να περνάει μέσα από μια απλοποιημένη διαδικασία. Οι εμπλεκόμενοι όμως ε, θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί μιλάμε για λίγα τέτοια προϊόντα ενώ τα νέα προϊόντα ε, δεν θα είναι κάποια προϊόντα που θα ωφεληθούν από τις διαδικασίες αυτές. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε μια, ένα ιστορικό ασφαλούς χρήσης. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στον τομέα της επιστημονικής παραγωγής γύρω από το ε, θέμα αυτό και απαιτείται μια πιο συγκεκριμένη διαδικασία για την δημιουργία ενός ιστορικού ασφαλούς χρήσεως. Γιατί αλλιώς θα είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατάει όσο κρατάει και η διαδικασία σήμερα για τα νέα προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν στο κόστος, μιλάμε για το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για να κάνει κανείς μια αίτηση για νέα προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί και από, την, από τον ξεκάθαρο χαρακτήρα των δηλώσεων της ΕΦΣΑ που θα κυκλοφορήσουν τον μήνα Οκτώβριο. ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μπορεί να συνεργαστούν για διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είναι πιο σύντομες εφόσον έχουν προηγηθεί αντίστοιχε στο παρελθόν. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων πάρα πολύ ισχυρές. Υπήρχαν ανησυχίες αυτή τη βιομηχανία ότι το καθεστώς της προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να χορηγηθεί, ιδιαίτερα όταν ένα πανεπιστημιακό όργανο παράγει δεδομένα, αναφέρονται τα δεδομένα αυτά σε μια επιστημονική δημοσίευση, οπότε δεν προστατεύονται τα στοιχεία αυτά και μπορεί να υποφεληθούν από αυτά διάφορες επιχειρήσεις παραγωγής, έρευνας κτλ είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου που είναι η προστασία των προϊόντων. Ευχαριστώ Στίβεν. Περνάμε τώρα στο ρόλο των εθνικών αρχών και των εθνικών υπηρεσιών και στα πλαίσια του συγκεντρωτικού συστήματος τα κράτη-μέλη και ο ρόλος τους θα είναι πιο περιορισμένος στα πλαίσια της αδειοποίησης για την κυκλοφορία νέων τροφίμων στην κοινοτική αγορά. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις και στα ερωτηματολόγια μάλλον λέγουν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθούν την ΕΦΣΑ να κάνει αξιολογήσεις ασφάλειας παρέχοντας την ε, εμπειρογνωμοσύνη τους και επηρεάζοντας έτσι τις αποφάσεις ε, στη φάση ε, της τελικής λήψης τους. Δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς την παρούσα φάση ε, το πόσο θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με παραδοσιακά προϊόντα που προέρχονται από άλλες χώρες. Αυτό εξαρτάται και από, το, την ποσότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους ε, υπεύθυνου για την ασφαλή κατανάλωση των προϊόντων. Τώρα, οι συστάσεις για το αν θα πρέπει να εμπλέκονται τα κράτη-μέλη στην ε, ε, διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας των νέων προϊόντων και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία του συγκεντρωτικού συστήματος. Υπάρχει ο κίνδυνος εδώ τα κράτη-μέλη να έχουν αντιρρήσεις σε πάρα πολύ τακτική φάση και αυτό θα αντισταθμιστεί από συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συλλαγωμένων δεδομένων. Και έτσι μόνο θα μπορέσουμε εμείς να διευκρινίσουμε καλύτερα την έννοια της ασφαλούς κατανάλωσης. Το τελευταίο ίσως σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε εξετάσει είναι η σχέση ανάμεσα στον προτινόμενο κανονισμό και στους υπόλοιπους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα. Αρκετά θέματα έχουν τεθεί εδώ από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας με τους οποίους συναντηθήκαμε και από πλευρά της ΕΦΣΑ επίσης για τα νέα προϊόντα τα οποία μπορεί να παρουσιάσουν ε, προβλήματα στην κατανάλωσή τους. μπορεί να απαιτηθεί η αξιολόγηση να γίνεται και από τον κανονισμό του 2006, τον 1924. Επίσης η επαλήθευση των ισχυρισμών για την τροφιμική αξία και τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει αποφυγή της επανάληψης αποστολής δεδομένων για τα συγκεκριμένα αυτά νέα προϊόντα και σε σχέση με τους ισχυρισμούς για, το, για τις επιπτώσεις στην υγεία. Πολλές φορές αυτά είναι καρπός κλινικών μελετών οι οποίες θα πετούν πάρα πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Αν αυτές οι διαφορετικού τύπου αξιολογήσεις γίνουν σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, τότε η περίοδος για την προστασία των δεδομένων δεν θα συμπέσει με την προβλεπόμενη και αυτό είναι προβληματικό για τις επιχειρήσεις και είναι ένα αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις να καταθέσουν αιτήσει για την τοποθέτηση νέων τροφίμων στην κοινοτική αγορά. Υπάρχει πάντα λοιπόν ο κίνδυνος επικάλυψης σχετικά με την αξιολόγηση των νέων τροφίμων που περιλαμβάνουν ε, θρεπτικές ουσίες ή ουσίες ε, για συγκεκριμένες δίαιτες και εδώ απαιτούνται διαφορετικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τον 609 του 2002. Υπάρχουν επιχειρήματα λοιπόν για τον συνδυασμό των δύο αυτών αξιολογήσεων σε μία μορφή αξιολόγησης έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, μη χρήσιμες επικαλύψεις. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε επίσης ιδιαίτερα από πλευρά των καταναλωτών είναι ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει εναρμόνιση σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το καθεστώς των πιθανών ε, ουσιών και συστατικών. Ε, μερικές ε, φυτικές ουσίες ε, μπορεί να θεωρούν τρόφιμα, θεωρούνται τρόφιμα σε ορισμένες χώρες, ενώ σε άλλες χώρες θεωρούνται φαρμακευτικές ουσίες και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο συγκεντρωτικό σύστημα. Γιατί οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μπορεί να καθυστερήσουν λόγω ακριβώς της διαδικασίας που ακολουθείται για τα νέα τρόφιμα τα οποία περιλαμβάνουν φυτικές ουσίες βότανα. Η πρόταση την οποία κάνουμε λοιπόν είναι ότι αν είναι δυνατόν οι αξιολογήσεις στον τομέα της ασφάλειας της κατανάλωσης και των ισχυρισμών για την υγεία να γίνονται ταυτόχρονα για την πενταετή περίοδο προστασίας που να ξεκινάνε δηλαδή την ίδια ημερομηνία και οι δύο διαδικασίες να λειτουργούν παράλληλα και όχι διαδοχικά η μία μετά την άλλη κάτι το οποίο θα αυξήσει τη χρονική προθεσμία, την ανάγκη για μια χρονική προθεσμία προστασίας των δεδομένων. Σχετικά τώρα με τις θρεπτικές ουσίες και τις ουσίες ε, συγκεκριμένης δίαιτας ε, θα πρέπει να μην, να μην ακολουθήσουν δύο διαφορετικές παράλληλες πορείες και περαιτέρω καθυστέρηση. Και τέλος η έλλειψη εναρμονισμού ε, σε σχέση με το καθεστώς ορισμένων βοτάνων και ορισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στα νέα τρόφιμα είναι θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της εναρμονισμένης ε, διακανονιστικής ε, ρύθμισης. Αυτά. Αυτό ήταν μια γενική περιγραφή λοιπόν της συμπληρωματικής μας αξιολόγησης. Εάν έχετε απορίες με τα χαράς να σας τις λύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγηση αυτή, την λεπτομερέστατη. Ευχαριστούμε και την Εύσα για την παρουσίασή της και θα δώσω τώρα το λόγο στον James Nicholson, ο οποίος είναι εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για τα νέα τρόφιμα. Ευχαριστώ και πρώτα να ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν ήμουν από την αρχή. Ε, έχω και άλλες υποχρεώσεις. Πάντως με την ευκαιρία ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσίαση ιδίως που τόνισε και ορισμένους τομείς ανησυχίας και οι σκιώδεις ηγητές και άλλοι συνάδελφοι μου τα έχουν πει αυτά να προσθέσω τώρα λίγα λόγια σύντομα για τρεις συστάσεις από τη μελέτη αντικτύπου όπου θα χρειαστούν σημαντικές τροποποίησεις μέσα από την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Πρώτα, ορισμός και πεδίο εφαρμογή της πρότασης που δεν έχει επιτύχει τους στόχους της να διευκρινίσει τον ορισμό των novel food και από τη μελέτη δικτύπου αλλά και από τις συζητήσεις που έχω κάνει εγώ φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει συνένεση σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του άρθρου 2 με τον ορισμό του novel food. Η αφαίρεση των κατηγοριών έχει οδηγήσει σε σημαντική ανησυχία στη βιομηχανία. Δέχομαι μεν ότι χρειάζεται κάποια ευκαμψία για να καλυφθούν κενά στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Παρ' όλα αυτά μου φαίνεται δύσκολο να δεχτώ την πρόταση της Κομισιόν που δεν έχει απολύτως καμιά ταξινόμηση μέσα. Είναι σημαντική συζήτηση βέβαια που την έχουμε κάνει και μέσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά και στο εργαστήρι Και σωστό είναι να επανισαχθούν οι κατηγορίες για να προληφθούν και κάποιες εξελίξεις από την πλευρά της βιομηχανίας. Σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων είναι κύριος στόχος της προτάσεως και το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίζει τα ιδιόκτητα δεδομένα από τα υπόλοιπα, αλλά βάζει και μια πενταετή περίοδο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες της βιομηχανίας, του κλάδου δηλαδή, για την προστασία δεδομένων και για τους ισχυρισμούς υγείας αλλά και για τους ισχυρισμούς θρεπτικής αξίας και ούτε να αποδειχθεί ότι μένει χωρίς καμιά αξία η περίοδος αδειοδότησης. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε την χρήσιμη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας μας και των επανεπιστημίων. Και είναι επίσης σημαντικό να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή, να μην περιοριστεί χωρίς λόγο από τους κανονισμούς Novel Food. Τώρα για τις προθεσμίες επανέρχομαι σε κάτι που λέει η μελέτη αντικτύπου που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα υπερβολικά πολλά στάδια της ε, διαδικασίας αδειοδοτήσεως. Εδώ πρέπει να γίνει ταχύτερη η διαδικασία αντιδοτήσεως για τα novel food. Πρέπει να επανεξετάσουμε να δούμε ξανά ποιοι είναι οι τομείς που πρέπει να επιβληθούν κάποιες προθεσμίες, να επιταχυνθεί όμως η διαδικασία και ο χρόνος που έχει στη διαθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκδώσει γνωμοδότηση πρέπει να μειωθεί από τους 9 μήνες καθώς και για την απόφαση της Διερκούς Επιτροπής. Αυτά ήθελα να πω για την ώρα, αγαπητέ Πρόεδρε. Θα επανέλθουμε. Θα ακούσω βέβαια και τους και ηγητές αλλά και άλλα μέλη και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, James. Ξεκινάμε με τους σκιώδεις, λοιπόν. Η κυρία Πιλάρα Γιούζο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον εισηγητή μας, ε, τους εκπροσώπους της ΕΦΣΑ και τους συντάκτες της γνωμοδότησης. Εμείς είχαμε, όπως είπατε, σε εκκρεμότητα το θέμα αυτό από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και ελπίζω να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από την εμπειρία που έχουμε σωρεύσει όλοι. Ήμασταν οι ίδιοι έτσι κι αλλιώς κάποιοι από μας ε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Σχετικά με την θέση του κυρίου Νίκολσον, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι οι ορισμοί. Οι ορισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, μας το είπαν αυτό οι εμπειρογνώμονες, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί η νομική ασφάλεια, η νομική βεβαιότητα σχετικά με, ε, με δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να κληθεί να χρησιμοποιήσουν και τις μεθόδους της νανοτεχνολογίας. Ε, πράγματι η πρόταση είναι αρκετά λογική, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι απαιτήσει στις διάφορες χώρες δεν συμπίπτουν μεταξύ τους σχετικά με την χρήση των τροφίμων και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για την προστασία των δεδομένων θα συμφωνήσω με αυτούς ε, που μίλησαν γύρω από το θέμα αυτό, ερευνητικές πανεπιστημιακές μονάδες ε, και πράγματι ε, πολλές φορές η βιομηχανία απαιτεί τα δεδομένα αυτά να είναι αποκλειστικής χρήσης και κάτι τέτοιο βέβαια δημιουργεί προβλήματα στα πανεπιστήμια και τα κέντρα ερευνών. Πολύ καλή ιδέα είναι αυτά τα οποία ακούστηκαν για τον τρόπο με τον οποίο θα κατατίθενται οι προτάσεις. Για την ΕΦΣΑ προφανώς θα πρέπει να συνεχίσει τις ε, δραστηριτές εργασίες της, θα πρέπει να λυθούν τα θέματα που αντιμετωπίζει ο εκπρόσωπος της ΕΦΣΑ. είπε ότι αυτό θα πρέπει να είναι δωρεάν, δεν θα πρέπει να ε, επιβάλλονται τέλη. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε εύκολα, δεν θα βρούμε εύκολα μια λύση στο πρόβλημα. Αυτό το οποίο ζητώ στην ΕΦΣΑ είναι να ξεκαθαρίσει και να δώσει συγκεκριμένες γραμμές στην βιομηχανία γιατί βλέπουμε ότι τώρα έχουμε πολύ συγκεκριμένα θέματα σε σχέση με το θέμα των ισχυρισμών στον τομέα της υγείας και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία. Σχετικά τώρα με τους άλλους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε να κάνουμε με κανονισμούς οι οποίοι προβλέπουν άλλα πράγματα διαφορετικά που ε, τώρα στις περιπτώσεις όπου υπάρχει η σύγχυση για τον χαρακτήρα των ουσιών, των συστατικών, θα πρέπει να υπάρξει ένας κανόνας έτσι ώστε να μην υπάρχουν δύο διαφορετικές χρονικές ε, περίοδοι προστασίας. Να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Τα νέα τρόφιμα τα οποία έχουν ήδη αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του κανονισμού του 2007 θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο κατάλογο. σε αυτή την περίπτωση δεν θα την χάνουν αυτής της προστασίας της οποίας πρέπει να την χάνουν ή ε, τα νέα τρόφιμα που έχουν αδειοδοτηθεί μέσα από τον καινούριο κανονισμό. Θα προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια βεταβατική περίοδο για να υπάρξει μια λύση σε σχέση με την χρήση και την κατανάλωση αυτών των προϊόντων και το, ε, την περίοδο πενταετούς προστασίας τους. Yes. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια για την αξιολόγηση. Εμείς οι πράσινοι έχουμε ακόμη το αίσθημα ότι τοποθετείτε τις επιχειρήσεις παραπάνω από τα συμφέροντα των καταναλωτών και την προστασία τους. Ενώ εμείς θα θέλαμε την πρώτη θέση να έχουν οι πολίτες και οι καταναλωτές και καταναλώτριες. Μετά για την πρόταση της Κομισιόν έχουμε μερικά σχόλια για τα κλωνοποιημένα τρόφιμα. Ανησυχούμε γιατί αποκλείονται από το εύρος της νομοθεσίας αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα καλύπτονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν τα κλωνοποιημένα τρόφιμα πριν εγκριθεί η νομοθεσία. Η ισχύουσα εθνική νομοθεσία δεν είναι τέλεια αλλά τουλάχιστον απαιτεί να υπάρχει διαδικασία διοδότησης πριν βγουν στην αγορά τα κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αν τα αποκλείσουμε από αυτή την νομοθεσία τότε θα μπορούσαν να μπουν στην αγορά αυτά τα τρόφιμα χωρίς να το καταλάβει κανείς. Για τα νανοσωματίδια Έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα του κατά πόσο θα πρέπει να πληροφορούνται οι καταναλωτές αν περιέχουν τέτοια σωματίδια τα τρόφιμα. Έχουμε ακόμη σοβαρές ανησυχίες. Όσο για τα όρια, εδώ γίνεται λόγος για τα νανοσωματίδια ως 50% ή παραπάνω σωματιδίων που φτάνουν μέχρι τα 100 Νανόμετρα. Νανόμετρα. Αλλά ακόμα και η ΕΦΣΑ αναγνωρίζει ότι δεν είναι ασφαλή και σίγουρα όλα αυτά και λέει το όριο να είναι 10%. Αν το 50% εφαρμοστεί, όχι μόνο για τις ετικέτες αλλά και για την ομοθεσία, για τον κανονισμό, τότε υπάρχει ο κίνδυνος μερικά νανοσωματίδια να μην καλύπτονται από τον ορισμό και άρα να μην θεωρούνται τμήμα των νέων τροφίμων. Άρα να μην γίνεται καμία τους αξιολόγηση. Τώρα για την αξιολόγηση του κινδύνου στην... πρέπει να έχουμε πιο συντηρητική αντιμετώπιση και να εφαρμόσουμε το όριο του 10% που συστήνει η ΕΦΣΑ. Τρίτον, για την εφαρμοστική πράξη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιες πράξεις για να καθοριστεί αν ένα τρόφιμο θεωρείται νέο ή όχι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν επέμενε ότι εδώ χρειάζονται κατεξουσιοδότηση πράξεις για τέτοια θέματα. Το ίδιο ισχύει και για την ενημέρωση του καταλόγου της Ένωσης. Γιατί τα νέα τρόφιμα να εγκρίνονται χωρίς να το εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ όλα τα άλλα πρόσθετα διατροφής εξετάζονται. Ακόμα και η παλαιότερη πρόταση του 8 της, Επιτροπής, Κομισιών έλεγε η ενημέρωση του καταλόγου να γίνει με την έγκριση του Κοινοβουλίου. Δεν είναι κατανοητό ότι τώρα η Κομισιόν προτείνει διαδικασία χωρίς το δικαίωμα του βέτο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Α, για μια στιγμή. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω την Επιτροπή, την ΕΦΣΑ και το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών. Σημερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τα γενετικά τροποποιημένα και τα κλωνοποιημένα προϊόντα που πρέπει να εξαιρεθούν από την πρόταση και πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μένουν σε εκκρεμότητα. Όταν εξετάζουμε επίσης ε, ε, τα παραδοσιακά λεγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες και σε σχέση με την ε, περίοδο την πενταετή θα πρέπει να τεθεί το θέμα προστασίας των προϊόντων αυτών ε, δεν ξέρω τι μεθόδους ακολουθούν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΦΣΑ για να ορίσουν ακριβώς τα κριτήρια ε, και τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται. Απαιτείται εδώ λοιπόν να ξεκαθαριστούν τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης τώρα, οι προτινόμενες αιτήσει δεν θα αποστέλλονται ξεχωριστά σε κάθε μία διαφορετική χώρα αλλά θα δίδονται απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΦΣΑ. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι αν κατάλαβα καλά να μειωθεί το χρονοβόρο της διαδικασίας αλλά ταυτόχρονα ε, δεν είναι τόσο ο χρόνος της διαδικασίας που παίζει ρόλο για αυτούς που εμπλέκονται αλλά η προβλεψιμότητα αν θέλετε της διαδικασίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μειώνεται ο ρόλος των κρατών μελών σχετικά με την χρήση των νέων προϊόντων, ιδιαίτερα όταν δεν γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΦΣΑ έχουν την δυνατότητα για να δώσουν τις απαιτούμενες διαβεβαιώσεις. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Μπόλεν. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Πότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, χθες ορίστηκα σκιοδησίτης για το θέμα από την ομάδα μου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έτσι είχα στη διάθεση μόνο χθε το απόγευμα για να εξετάσω τη μελέτη αντικτύπου. Ομολογώ ότι μένω εμβρόντιτος το ίδιο, όπως και πέρσι, που είχα λάβει τον φάκελο ERM, από την πρόταση. Τι πρόταση είναι αυτή εδώ, πρέπει να αλλάξουμε ήδη τους ορισμούς για να είναι πλέον σαφές τι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για να ξεκαθαρίσουμε περί τίνος πρόκειται, για να υπάρχει κάποια λογική. Και εγώ τώρα πώς να τοποθετηθώ απέναντι στην πρόταση όταν οι ίδιοι εμπειρογνώμονες λένε ότι εκατοντάδες χιλιάδες τρόφιμα έχουν προκύψει και χαρακτηρίζονται ως νέα τρόφιμα από το 1997 και μετά. Βλέπω λοιπόν εδώ πέρα μεγάλο βαθμό ανασφάλειας. Και για την ίδρυση αυτή του κεντρικού φορέα που αφενός υπάρχουν ανησυχίες ότι θα επιβαρυνθεί υπερβολικά το έργο του. Από την άλλη μεριά υπάρχει φόβος ότι ενδέχεται ορισμένες επικίνδυνες ουσίες να μην εμπίπτουν καν στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Ε, ε, επαναλαμβάνω ότι έχω μείνει πραγματικά άναυδος. Ελπίζω ότι η συνεργασία με τον κύριο Νίκολσον θα οδηγήσει στο τουλάχιστον αυτή η μεγάλη ε, έκπληξή μου να ε, οδηγήσει σε κάποια θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. που βάλατε το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ και για την Επιτροπή σας που έδειξε ενδιαφέρον της ε, για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή και τον εισηγητή Νίκολσον γιατί προσπάθησαν να προχωρήσουν σε ένα θέμα περίπλοκο και προσπάθησαν να βρουν μια κάποια ισορροπημένη διατύπωση μετά από τις αρνητικές εμπειρίες του 2009-2010 που μας είχαν οδηγήσει εκείνη την εποχή ε, να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε ε, σε λεπτομέρειες το σύνολο του πακέτου χωρίς όμως να το ολοκληρώσουμε. Ε, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση που προηγήθηκε ιδιαίτερα υπό το φως ε, της ε, νέας προσπάθειας που θα κάνει η Ιταλική Προεδρία και υπό το φως μιας πιθανής συμφωνίας η οποία ελπίζουμε να ε, ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν από τα θεσμικά όργανα. Από πλευράς του Συμβουλίου Υπουργών αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η Ελληνική Προεδρία ήδη είχε θέσει προσυζήτηση επανειλημμένα το θέμα και μετά από τις προσπάθειες αυτές τώρα εναπόκειται στην Ιταλική Προεδρία να ορίσει κάπως περισσότερο τα θέματα τα οποία παραμένουν ε, ε, σε εκκρεμότητα. Αναφέρομαι εδώ στον, στη μορφή που θα πρέπει να πάρει ο κατάλογος των νέων τροφίμων και ο, καθορισμός, ο ορισμός επίσης ε, του τι είναι νανοηλικό. Από πλευράς μας είμαστε διατεθειμένοι το ταχύτερο δυνατόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, όντας βέβαια όσο επιφυλακτική χρειάζεται, όντας όσο προσεκτική χρειάζεται λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος. Μπορούμε να πούμε πάντως από τώρα ότι θα δώσουμε κάθε δυνατή προσοχή σε όλες τις απόψεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί από πλευράς ε, των ε, ε, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Λοιπόν, η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από πλευράς μας θα γίνει και ταυτόχρονα θέλουμε να συνεργαστούμε εφόλης της ύλης με το Κοινοβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει για μας ένα σημαντικότατο σημείο αναφοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ιταλική Προεδρία. Δεν ξέρω τώρα αν οι εμπειρογνώμονες θέλουν να επανέλθουν και να προσθέσουν κάτι ή να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα σχόλια τα οποία προηγήθηκαν. Αν υπάρχει, όχι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και γι' αυτό θα δώσω το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στον εισηγητή μας για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης για την χρήσιμη συζήτηση. Για τον ορισμό πρώτα, δεν είναι πρόθεση της Κομισιόν να περιλάβει novel food σε αυτόν τον ορισμό που δεν θεωρήθηκε novel food στο παρελθόν. Όπως είπα και εισαγωγικά, υπήρξε αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής. Εμείς επιθυμούμε να διασαφίσουμε τον ορισμό έτσι ώστε να λειτουργήσει και υπέρ των καταναλωτών και υπέρ των βιομηχανιών, να έχουν δηλαδή την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου, να γνωρίζουν και οι δύο πλευρές τι είναι νόβελ και τι όχι. Δεν είναι πρόθεσή μας λοιπόν να καλύψουμε αναδρομικά ή αδίποτε τρόφιμα τα οποία δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται novel food, αλλά να διευκρινίσουμε τις κατηγορίες. Παράδειγμα, υπό τον υφιστάμενο κανονισμό, για παράδειγμα, πρωτεΐνες που παράγονται από έντομα θεωρούνται novel food. Το έντομο όμως το σύνολό του δεν είναι novel food. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό και αυτό, σε αυτό μάλλον ευθύνεται ο ορισμός της οδηγίας που λέει προϊόντα τα οποία παράγονται από κάτι άλλο. Αυτή είναι η δυσκολία. Η πρόθεση λοιπόν των νομοθετών τότε ήταν αυτή. Βεβαίως εμείς είμαστε διατεθειμένες να βελτιώσουμε, να συμβάλλουμε στη βελτίωση του ορισμού του πεδίου εφαρμογή και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Για τον κατάλογο, για τη λίστα. Θα υπάρχει ένας ενιαίος κατάλογος και αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι ότι πολλά τρόφιμα υπόκειται στην substantial equivalence. Όταν δηλαδή κάποιος έχει λάβει άδεια υπάρχουν και άλλοι και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν αγορά παρόμοια τρόφιμα ή τα ίδια τρόφιμα διότι έχουν την ουσιώδη αυτή ισοδυναμία. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να μπει στη λίστα όταν θα ισχύσει ο νέος κανονισμός και όλα τα ε, προηγούμενα να θεωρηθούν ως generic χωρίς εμπορική επωνυμία. Αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσει να ισχύσει και η ε, ρήτρα περί ουσιώδους ισοδυναμίας. Ε, σας βεβαιώνω επίσης ότι τρόφιμα από κλόνους αποκλείονται διότι δεχθήκαμε όταν αρχίσαμε να κάνουμε την πρόταση ότι τρόφιμα από καθορίζονται σε ξεχωριστή νομοθεσία. Αν βέβαια η ξεχωριστή νομοθεσία δεν εγκριθεί ταυτόχρονα με τούτην εδώ, τότε τα τρόφιμα από κλόνους θα τα διατηρήσουμε μέσα στο πεδίο εφαρμογή της παρούσας οδηγία, ώστε να μην υπάρξει νομικό κενό βεβαίω δεν έχει ζητηθεί να περάσουν τα τρόφιμα αυτά στην αγορά αλλά όσο δεν υπάρχει ακόμα η άλλη νομοθεσία για την κλωνοποίηση θα κάνουμε αυτό. Τα GMO πάντοτε αποκλείστηκαν από τον κανονισμό και θα παραμείνουν ένα αποκλεισμό γιατί τα καλύπτουν άλλα νομοθετήματα για τα νάνο θεωρούμε σωστό και για την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και για τις βιομηχανίες να αναφερθούμε σε έναν υφιστάμενο ορισμό έστω και αν υπάρχει μοναχά για λόγους επισημάνσεως γιατί είναι πολύ τεχνικός και επιστημονικός ορισμός αυτός από μόνος του και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε κιόλα. γιατί έτσι είναι τα νανοηλικά. Βρίσκουμε λοιπόν πολύ σημαντικό να μην έχουμε ξεχωριστούς ορισμούς σε ένα ενίο τομέα, δηλαδή των τροφίμων, για τα νανοηλικά και είναι σημαντικό να παραμείνουμε όσο πιο συνεκτικές γίνεται με τους τεχνικούς ορισμούς της νομοθεσίας. Αν υπάρχουν βέβαια κάποιες ελαφρές διαφορές θα δούμε, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλους και για τους καταναλωτάς και καταναλωτρίας και για τις επιχειρήσεις. Βέβαια η ευρωγνωμοσύνη των χωρών μελών όπως εξήγησε και η Εύσα προηγουμένως θα παραμείνει Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει ε, να απλουστευτεί και η ΕΦΣΑ και για άλλους φακέλους συνεργάζεται στενά με τις χώρες και με τους επιστημονικούς οργανισμούς των και για τους χειρισμούς υγείας και τα νέα τρόφιμα είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι η νομοθεσία περί χειρισμών υγείας αναφέρεται στο εάν ένα τρόφιμο μπορεί να ισχυριστεί ο παραγωγό ότι είναι καλό για τα κόκαλα, για την καρδιά ή για πρόληψη ασθενειών. Αυτή η χειρισμοί υγείας, η σχετική νομοθεσία δηλαδή, εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα. Δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τα novel food. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτή η νομοθεσία να υπάρχει ξεχωριστά και όταν τυχαίνει να εφαρμόζεται σε novel food, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η νομοθεσία αυτή αναφέρεται στην ασφάλεια του τροφίμου, ενώ ο ισχυρισμό υγεία στην αποτελεσματικότητα της, του ισχυρισμού. Δηλαδή, αν όντω πραγματικά ε, προσφέρει κάτι στα κόκκαλα στην καρδιά κλπ. Άλλο λοιπόν είναι η νομοθεσία αυτή που πρέπει να λέει ότι είναι ασφαλές το novel food. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή αυτέ οι δύο νομοθεσίε να εφαρμόζονται εκ παραλίλου, μπορεί να είναι και διαδοχικά. Νομίζω ότι συμφωνούμε, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη του διαφορετικού αυτού στόχου των νομοθετημάτων. Σα ευχαριστώ και πάλι για τη χρήσιμη συζήτηση. βεβαίω θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μα και με το Συμβούλιο των Υπουργών και με την συνέλευσή σας και ίσως καταφέρουμε να εγκριθεί και σε πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε Κομισιόν. Και τώρα για να καταλήξουμε εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους όσους ε, λάβαν το λόγο. Ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση σήμερα και ελπίζω να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Σας διαβεβαιώνω ότι για μένα τα νέα τρόφιμα με ενδιαφέρουν, όχι τα κλωνοποιημένα. Αυτό είναι άλλο θέμα, χωριστό. Δεν σκοπεύω λοιπόν να μπερδευτώ με αυτό το θέμα των κλωνοποιημένων. Άλλοι θα ασχοληθούν. Θα κάνω μια ενημέρωση και θα σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα την επόμενη φορά και ελπίζω στο εργαστήριό μας της 7 Οκτωβρίου να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Δύο-τρία λεπτά έχουμε ακόμα. Σας υπενθυμίζω ότι στις παρατέταρτο, τρεις παρατέταρτο θα γίνει η οικογενειακή φωτογραφία. Σας κατευχαριστώ.